Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε την συνεδρίαση της Επιτροπής μας, ελέγχου του προϋπολογισμού. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχουν προτάσεις αλλαγής στην ημερησία διάταξη. Σας υπενθυμίζω ότι βρισκόμαστε και σε εκπομπή στο διαδίκτυο. και θα εξετάσουμε σήμερα τη διαδικασία απαλλαγής για το 2012. Χαίρομαι για την παρουσία του ε, κυρίου Σταϊκούρα ως εκπροσώπου του Συμβουλίου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας κυρίου Σταϊκούρα. Υπήρξε μια θέση που, μια σύσταση που έχει υπάρξει από την πλευρά του Συμβουλίου για τη διαδικασία αυτή της ε, απαλλαγής. Υπάρχει συμφωνία για το θέμα αυτό και θα θέλαμε να συζητήσουμε με το θέμα αυτό της απαλλαγής με τον κύριο Σταϊκούρα. Είναι γνωστό ότι 80% του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται σε διαμεμερασμένη αρμοδιότητα, επομένως συνδιαχείριση με τα κράτη-μέλη και ιδίως ε, και με περιφερειακές αρχές των κρατών μελών και όχι μόνο εθνικέ, παίζουν τα κράτη-μέλη ένα σημαντικό ρόλο επομένω, για το εγχείρημα μια βελτιότερης διαχείριση του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση, και όταν το Ελεκτικό Συνέδριο παρατηρεί ότι υπάρχει αύξηση των σφαλμάτων σε ορισμένου τομεί, παραδείγματο χάρη για την αγροτική ανάπτυξη, τα κονδύλια αγροτική ανάπτυξη, είναι τότε πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε και στον χώρο των κρατών μελών να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την παρουσία σας σήμερα ως εκπροσώπου της Προεδρίας του Συμβουλίου και για το γεγονός ότι έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις μαζί σας ως εκπροσώπου του Συμβουλίου και γνωρίζουμε ότι φυσικά το Συμβούλιο δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για μεμονωμένα κράτη-μέλη γιατί το κάθε κράτος μέλος έχει τη δική του νομοθετική αυτονομία, αλλά φυσικά και εσείς εκπροσωπείτε μια περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης θέλω να χαιρετήσω και πάλι τον κύριο Σεμέτα, ο οποίος έρχεται ενώπιον μας ως εκπρόσωπος της ε, Κομισιόν. Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι η Κομισιόν μας δίδει τακτικά αναφορές για τα θέματα αυτά και φυσικά θεωρούμε ότι και εμείς έχουμε καθήκον να ελέγχουμε την Κομισιόν και να υποβάλουμε προτάσεις για βελτίωση των ε, συνθήκων στα θέματα αυτά ελέγχου του προϋπολογισμού και η Κομισιόν φυσικά ε, πολλές φορές ακούει από εμά και από την κοινή γνώμη προτάσεις και επικρίσεις για θέματα τα οποία δεν μπορεί να επηρεάσει άμεσα αλλά μόνο έμεσα. Ένα θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει επίσης είναι το θέμα της ε, απαλλαγής του Συμβουλίου εδώ μπορεί να έχει κανείς διαφορετικές απόψεις για επιμέρους σημεία αυτής της διαδικασίας απαλλαγής και το κατανοούμε αυτό. Εγώ μπορώ απλώς να παρουσιάσω την άποψη της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Ο αρμόδιος συζητητής, ο κ. Σίβαν, δεν είναι παρόν σήμερα, αλλά το συζητήσαμε το θέμα αυτό αυτή την εβδομάδα και η άποψή μας είναι ότι και ο προϋπολογισμός του Συμβουλίου θα πρέπει να υπόκειται σε μια διαδικασία απαλλαγής δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν προϋπολογισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίοι δεν υπόκεινται σε έλεγχο από άμεσα εκλεγμένα κοινοβούλια. Τουλάχιστον θα πρέπει να μπορούμε να θέσουμε ερωτήσεις για αυτό το προϋπολογισμό του Συμβουλίου. Το γνωρίζει και ο, ο κύριος Υπουργός. Απλώς θέλω να υπενθυμίσω την στάση της Επιτροπής μας για τα θέματα αυτά και να την επιβεβαιώσω. Η Ελληνική Προεδρία, αγαπητοί συνάδελφοι, έχει αναλάβει τα ηνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δύσκολους καιρούς. Κύριε Σταϊκούρα, χαιρόμαστε πάρα πολύ για το γεγονός ότι η χώρα σας, η Ελλάδα, έχει θετικά οικονομικά αποτελέσματα να παρουσιάσει μετά από πολλά χρόνια δυσκολίας που οδήγησαν σε πολύ δύσκολες και οδυνηρές συνθήκες για τους πολίτες της, Ευρώπη, της Συγγνώμη. Έχουμε συζητήσει για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Τρόικα και το ποια μέτρα ήταν απαραίτητα και εύλογα. Πιστεύει η Επιτροπή μας όμως ότι ένας καλός δημοσιονομικός έλεγχος σε όλα τα κράτη-μέλη μπορεί να δράσει άμεσα και αποτελεσματικά στο να αποφευχθούν οικονομικές κρίσεις στο μέλλον και φυσικά και ο, ο δημοσιονομικός έλεγχος είναι τμήμα του δημοκρατικού ελέγχου και όταν λειτουργεί σωστά μπορεί να μας προστατεύσει από αρνητικές εξελίξεις όπως είναι η υπερχρέωση ενός κράτους. Καλώς ήλθατε λοιπόν και θα ήθελα να σας δώσω το λόγο κύριε Υπουργέ. Χαιρόμαστε λοιπόν που είστε εδώ και έχετε το λόγο. Mr. President. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Επίτροπε Σαμέτα, κυρίε και κύριοι. Είναι μεγάλη τιμή για μένα ε, η παρουσίαση των συστάσεων του Συμβουλίου για την απαλλαγή προς την Επιτροπή για την εφαρμογή του ενωσιακού προπολογισμού για το οικονομικό έτος 2012. Το θέμα είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα και λογοδοσία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Διαχείρισης για την εφαρμογή του προϋπολογισμού. Το Συμβούλιο αποδίδει πρωταρχική σημασία στη χρηστή οικονομική διαχείριση των ενωσιακών πόρων. Γι' αυτό εξέτασε λεπτομερώς τους τελευταίους μήνες την εφαρμογή του Προϋπολογισμού για το 2012 στη βάση της ετήσια έκθεσης του Ελεκτικού Συνεδρίου και της ε, δήλωσης αξιοπιστίας. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ε, στα πλαίσια της επικοδομητικής συνεργασίας με τα κράτη-μέλη είναι μια αυστηρή, ένα αυστηρό και πολύ ισορροπημένο κείμενο που ταυτοποιεί προβλήματα και προτείνει κατευθυντήριες γραμμές. Το έγγραφο αυτό, η σύσταση, υιοθετήθηκε την Τρίτη από το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ και σας το παρουσιάζω σήμερα στην Επιτροπή σας. Το ΕΚΟΦΗΝ επίσης υιοθέτησε συστάσεις για τις αποκεντρωμένες ε, υπηρεσίες και οργανισμούς, τους εκτελεστικούς οργανισμούς και τις κοινέ προσπάθειες. Με αυτόν τον τρόπο το Συμβούλιο επαναβεβαιώνει ότι υπάρχουν μια σειρά στοιχεία, κατά τη γνώμη του, όπου θα πρέπει να υπάρξει συνέχεια και εφαρμογή αυτών που προτείνει από την Επιτροπή και τους οργανισμούς ε, χωρίς καθυστέρηση. Στα πλαίσια αυτά το Συμβούλιο επίσης επαναβεβαίωσε την επιθυμία του να υπάρξει κάθε χρόνο πρόοδος στα συστήματα οικονομικής διαχείρισης και για να μειωθούν τα ποσοστά σφαλμάτων για τις πληρωμές στον προπολογισμό. Ιδιαίτερα, όπως είπε ο Πρόεδρος, επειδή ε, τα ποσοστά σφαλμάτων παραμένουν πάνω από το όριο σημαντικότητας και αυξήθηκαν το 2009. Παρά το γεγονός ότι είναι λιγότερα από την περίοδο πριν το 2009, και επειδή επίσης και παρά το ότι ένα τμήμα της αύξησης οφείλεται σε αλλαγή της ε, μεθοδολογίας ε, δειγματοληψίας του ηλεκτρικού συνεδρίου. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα αποτελέσματα, παρακαλώ επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας τις, τα βασικά πορίσματα των συστάσεων του Συμβουλίου. Πρώτα απ' όλα, το Συμβούλιο καλωσορίζει την ανεπιφύλακτη γνώμη του συνεδρίου για την αξιοπιστία των ετησίων λογαριασμών για τις υποχρεώσεις και για τα έσοδα και τις διοικητικές δαπάνες. Ωστόσο, το Συμβούλιο ανησυχεί διότι οι λειτουργικές δαπάνες ακόμη παρουσιάζουν λάθη επί ουσία και ότι σημαντικοί τομεί πολιτικής όπως η ανάπτυξη της υπαίθρου, η συνοχή και η έρευνα παρουσιάζουν μεγάλο ποσοστό σφαλμάτων. Παράλληλα, το Συμβούλιο σημειώνει ότι όπως και προηγούμενα χρόνια, τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου είναι μόνο εν μέρει αποτελεσματικά για να διασφαλίζουν την νομιμότητα και κανονικότητα των δοσοληψιών. Το Συμβούλιο γνωρίζει ότι η καλύτερη δαπάνηση και η χρηστή οικονομική διαχείριση των πόρων έχει ιδιαίτερη σημασία για το πώς αντιμετωπίζει η κοινή γνώμη τις δράσει που χρηματοδοτούνται από τον ενωσιακό προπολογισμό. Οπότε, το Συμβούλιο στηρίζει σταθερά τις συστάσεις που υπέβαλε το συνέδριο και επιμένει ότι πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως. Στις συστάσεις του, το Συμβούλιο εκφράζει την απογοήτευσή του για τα αποτελέσματα των ελέγχων για την ανάπτυξη της υπαίθρου, διότι το ποσοστό σφαλμάτων παραμένει υψηλό. Παράλληλα, το ποσοστό σφαλμάτων για την περιφερειακή πολιτική εξακολουθεί να είναι σε σχετικά υψηλό επίπεδο. Στα πλαίσια αυτά το Συμβούλιο επαναβεβαιώνει την ανάγκη η Κομισιόν να ενισχύσει τη συνεργασία της με τα κράτη-μέλη με στόχο να υπάρξει πιο στοχευμένη βοήθεια ούτως ώστε οι έλεγχοι να είναι πιο αποτελεσματική και να εφαρμόσουν όλα τα αναγκαία προληπτικά και διορθωτικά μέτρα. Περαιτέρω, το Συμβούλιο σημειώνει σε σχέση με τις παρατηρήσεις του συνεδρίου ότι ένα σημαντικό τμήμα των ε, πράξεων που παρουσίασαν λάθη, για ένα τέτοιο σημαντικό τμήμα, οι εθνικές αρχές είχαν αρκετή πληροφόρηση για να εξεύρουν και να διορθώσουν τα λάθη. Οπότε το Συμβούλιο τονίζει ότι ε, αποτελεσματικές δομές ε, διοικητικές και ελέγχου ε, συμπεριλαμβανομένης και μιας αξιόπιστης δυνατότητας ελέγχου είναι στοιχεία κλειδιά για να διορθώνονται και να, μάλλον για να ε, προλαμβάνονται τα λάθη και καλεί την Κομισιόν να ενισχύσει να ασκεί πλήρω τον ε, εποπτικό ρόλο της ούτως ώστε να υπάρχει ουσιαστική προστασία του ενωσιακού προπολογισμού. Θέλω να είμαι σαφής από αυτού. Βεβαίως, οι βελτιώσεις ε, θέλουν χρόνο για να καταστούν ε, σαφείς, λαμβάνοντα υπόψη και το περίπλοκο νομικό πλαίσιο σε σχέση με τις ενωσιακές δαπάνε η απλούστευση και εναρμόνιση των κανόνων και των συνθήκων ε, επιλεξιμότητας είναι θεμελιώδους σημασίας για να επιτευχθεί μία ε, ανεπιφύλακτη γνώμη κατά τον έλεγχο. Η υιοθέτηση ε, των νέων νομοθετημάτων που εφαρμόζουν το νέο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και ο νέο δημοσιονομικό κανονισμός περιέχουν νέα και συμπληρωματικά στοιχεία ελέγχου και υποχρεώσεις εκθέσεων. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία για να επιτευχθεί σημαντική πρόοδος προς την απλούστευση, τη διευκρίνηση και την συνέπεια των κανόνων, ούτω ώστε να αυξηθεί η συμμόρφωση. Έχουμε διάφορα νέα όργανα δυνατότητε, όπω οι απλουστευμένε δυνατότητε για το κόστο, που ήδη εφαρμόζονται από την Κομισιόν. Παράλληλα, πολλά πρέπει ακόμη να γίνουν στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων ιδιαίτερα σε τομείς ε, επιμερισμένης διαχείρισης, όπου οι εθνικοί κανόνες ε, στα κράτη-μέλη εφαρμόζονται ακόμη. Ο εξυγχρονισμός και η απλούστευση των διαδικασιών δημοσίων προμηθειών πρέπει λοιπόν να συνεχιστεί. Το Συμβούλιο ενθαρρύνει την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη να εναρμονίσουν περαιτέρω τους κανόνες τους, ούτως ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος λαθών. Ένα απλούστερο κανονιστικό πλαίσιο σε συνδυασμό με καλύτερη βοήθεια προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς θα μας βοηθήσει να έχουμε μια πιο αποτελεσματική και διαφανή διαχείριση των ενωσιακών πόρων. Κυρίε και κύριοι, στην ετήσια έκθεσή του για το 2012 το συνέδριο αφιέρωσε ιδιαίτερη προσοχή στις ε, οικονομικές διορθώσεις και τους μηχανισμούς ανάκτησης. Κατά τη γνώμη του Συμβουλίου, πρόκειται για πολύ σημαντικά εργαλεία για την μακροπρόθεσμη προστασία του νοσιακού προπολογισμού. Το Συμβούλιο λοιπόν καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει όπου χρειάζεται την εφαρμογή όλων των διαθέσιμων διορθωτικών μέτρων. Η αυστηρή εφαρμογή αυτών των μηχανισμών θα βελτιώσει την ε, διαχείριση των πόρων, θα αυξήσει τη διαφάνεια και θα βελτιώσει τα θετικά αποτελέσματα που προκύπτουν από την ε, δαπάνη ενωσιακών πόρων για την Ευρώπη. Βεβαίως πρέπει να τονίσουμε ότι είχαμε 4,4 δισεκατομμύρια οικονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις το 2012 που είναι τριπλασιασμό σε σχέση με το 2011. Αυτό είναι θετικό αποτέλεσμα προς την ίδια Αυτό αποτελεί 3,2% των συνολικών πληρωμών για το 2012. Ενώ ο μέσος όρος για την περίοδο 2019-2012 ήταν 2%. Ανάλογα με το σχέδιο έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωστόσο, η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη από τη θεραπεία. Γι' αυτό το Συμβούλιο καλεί την Κομισιόν να συνεχίσει την αυστηρή εφαρμογή όλων των διαθέσιμων προληπτικών μέτρων και να εφαρμόσει αυστηρά και πλήρως σύμφωνα με τους ε, κανόνες τη διακοπή και αναστολή ε, πληρωμών, ούτω ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι για την νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων. Κυρίε και κύριοι, να στραφώ τώρα στα εσωτερικά συστήματα διαχείριση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Συμβούλιο θεωρεί ότι η ετήσια έκθεση δράση που έχουν ε, εκπονήσει οι Γενικοί Διευθυντέ Κομισιών και οι παρατηρήσει που περιέχονται σε αυτέ τι εκθέσει είναι σημαντικά και χρήσιμα έγγραφα που ε, επιτρέπουν να υπάρχει διαφάνεια και λογοδοσία στα κράτη-μέλη και στο κοινό. Οι παρατηρήσεις λοιπόν θα πρέπει να εφαρμόζονται συστηματικά όποτε είναι σκόπιμο για να βελτιωθεί η αξία αυτών των εκθέσεων. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι το Συμβούλιο εκτιμά την εργασία του συνεδρίου στην προσπάθεια αποτίμησης των αποτελεσμάτων που επιτυχάνονται από τον ενωσιακό προπολογισμό. Περαιτέρω, υπό το φως ε, της αύξησης των υπολείπων προς εκαθάριση ή των εκκρεμούσων ε, υποχρεώσεων, το ε, συνέδριο καλεί την Κομισιόν να προετοιμάσει και να δημοσιεύσει μία πρόβλεψη μακροπρόθεσμη για τις ταμιακές ζωές που να προσπαθεί να προβλέψει τις μελλοντικέ ανάγκες πληρωμών για να καθορίσουμε τις μελλοντικέ ανάγκες, να προγραμματίσουμε καλύτερα τις ε, δημοσιονομικές προτεραιότητες και να διασφαλίσουμε ότι οι αναγκαίες πληρωμές μπορούν να γίνουν από τους εγκεκριμένους ετήσιους προϋπολογισμούς. Προς την κατεύθυνση αυτή το Συμβούλιο συμφωνεί με το συνέδριο ότι πρέπει να ε, προχωρήσουμε πέρα από μια πολιτική που βασίζεται στη συμμόρφωση και να εστιάσουμε στην απόδοση. Αυτό σημαίνει, πως αυτό σημαίνει πως πρέπει να έχουμε ρωμαλαίους μηχανισμούς, ούτως ώστε να έχουμε έγκαιρα, αξιόπιστα και συγκρίσιμα στοιχεία για να μπορούμε να μετρήσουμε και να κάνουμε απολογισμό για την απόδοση. Το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο μπορεί μέσω των νέων ε, μηχανισμών μηχανισμών που προβλέπει να διασφαλίσει ότι θα πρέπει να είναι σαφές το όφελος από την εφαρμογή των νοσιακών πολιτικών. Κυρίε και κύριοι, όλες αυτές οι σκέψεις και οι προτάσεις οδήγησαν το Συμβούλιο Κοφίν να προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να χορηγήσει απαλλαγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή του Γενικού Προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ για την παρουσίασή σας. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εισηγητή μας Μάρκος Μπίμπα, αλλά ίσως η Κομισιόν θέλει πρώτα να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι. Χαιρετίζω αυτά τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που είναι τόσο ισορροπημένα και την Ελληνική Προεδρία για όσα έκανε για το θέμα αυτό των απαλλαγών. Όπως είπα και την Τρίτη στο ΕΚΟΦΗΝ, η Κομισιόν θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη για να εφαρμόσουν σωστά τα προγράμματά τους και να χρησιμοποιήσουν πλήρως όλα τα μέτρα που προβλέπει το δημοσιονομικό πλαίσιο μέχρι το 20 για να μειωθεί ο κίνδυνος λαθών. Ιδιαίτερα τονίζουμε προς τα κράτη-μέλη ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουν την απλοποίηση των κανόνων και διαδικασιών και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Πράγμα που θα βοηθήσει την καλύτερη εφαρμογή και το λιγότερο κόστος και επίσης τη μείωση του κινδύνου λαθών. Η Κομισιόν βέβαια θα τονίσει τις ε, εποπτικές της ε, δραστηριότητες και με προληπτικό τρόπο και με διορθωτικό όπου το ελεκτικό συνέδριο έχει ταυτίσει λάθη. Αλλά οι πραγματικές αλλαγές θα εφαρμοστούν μόνο όταν τα κράτη-μέλη αναλάβουν τις ευθύνες τους όταν μιλά, ε, μιλώντας για θέματα διαχείρισης κοινή. Η πρόληψη βέβαια είναι πάντα καλύτερη από τη θεραπεία και αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο όταν μιλάμε για την πρόληψη λαθών για κοινοτικά κονδύλια και πόρους. Και τα εθνικά προγράμματα πρέπει επίσης να είναι αποτελεσματικά για τους πολίτες. Αυτή τη στιγμή γίνονται πολλά για να εφαρμοστεί το νέο πλαίσιο αποτελεσματικότητας για να υπάρξει καλύτερη εποπτεία της προόδου και των αποτελεσμάτων όλων των προγραμμάτων. Το άρθρο 318 ή η έκθεση μάλλον αποτίμησης με βάση το 318 θα είναι ένα πολύ σημαντικό έγγραφο που θα υποβάλουμε και θα το βελτιώσουμε και εμείς. Τέλος, οι τρεις χώρες μέλη που δεν ε, ε, ενέκριναν την απαλλαγή. Δεν βλέπω καμία διαφορά μεταξύ αυτών που λέει η κοινή δήλωση και αυτών που λέει το Συμβούλιο. Όλες και οι τρεις συμφωνούν ότι πρέπει από κοινού να διορθωθούν τα λάθη και να γίνουν περισσότερες προσπάθειες. Και αυτό σημαίνει ιδιαίτερα τα κράτη-μέλη που έχουν την πρώτη ευθύνη για 80% της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Να μην ξεχνάμε ότι έχουν βρεθεί λάθη μόνο σε εθνικό επίπεδο και η Κομισιόν απέδειξε ότι μπορεί και έχει προστατεύσει τα οικονομικά, τους οικονομικούς πόρους της Ένωσης αποτελεσματικά και έχει ζητήσει επανειλημμένως από τα κράτη-μέλη να ε, είναι περισσότερο υπεύθυνα και να έχουν περισσότερη λογοδοσία οι εθνικές δηλώσεις θα συζητηθούν από την Κομισιόν αλλά πρέπει να όλοι οι παράγοντες που πρέπει να πετύχουν τη διαφάνεια να τις εφαρμόσουν. Γι' αυτό δεν δεχόμαστε τη συστάση των τριών αυτών χωρών και ελπίζω να δεχτούν τελικά την εγγύηση που δίνει η Κομισιόν για την ε, σωστή διαχείριση των πόρων της Ένωσης και εθνικά και ενωσιακά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Επιτροπέ. Αρχίζει τώρα η συζήτηση. Πρώτα πρώτα ο εισηγητής μας. Ο κύριος Πίπερ, ο εισηγητής μας έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, Θέλω να θέσω ένα ερώτημα στον κύριο Τόιερ, στον πρόεδρό μας για την ημερήσια διάταξη προηγουμένως. Ναι. Προφανώς ο κύριος Επίτροπος έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα για τα θέματα τα συνολικά της ε, απαλλαγής αλλά θα ήθελα να σταθώ τώρα στο θέμα της παρουσίασης του, της Προεδρίας του Συμβουλίου. Θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τα λόγια σας. Θέλω και εγώ να σας εκφράσω την προσωπική μου ευγνωμοσύνη για τη διαδικασία μεταρρυθμίσεων που έχει περάσει η χώρα σας και συνεχίζει φυσικά και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στα εγχειρήματα αυτά. Σε ό,τι αφορά το ίδιο το Συμβούλιο των Υπουργών και τη θέση του Συμβουλίου, είμαι κάπως διχασμένος σε σχέση με τα συναισθήματά μου. Έχω από τη μία πλευρά την εντύπωση ότι το Συμβούλιο μας ζητά να δώσουμε την απαλλαγή και εδώ υπήρξε κάποια πίεση από ό,τι φαίνεται από ορισμένες, χώρες, στο Συμβούλιο. Υπάρχουν αυτές οι τρεις χώρες οι οποίες δεν υποστηρίζουν τη θέση του Συμβουλίου είναι η Σουηδία, οι κάτω χώρες και η ε, Ολλανδία, ή το Ηνωμένο Βασίλειο. Και φαίνεται να μην συμφωνούν με αυτά που μας έχετε παρουσιάσει σήμερα εδώ. Και γι' αυτό είμαι υποχρεωμένος να θέσω κάποιες κάπως δυσάρεστες ερωτήσεις Αναφερθήκατε στην ε, διαδικασία απαλλαγή και έχετε ε, επενέσει τις διαδικασίες δημοσιονομικών διορθώσεων που επήλθαν στο 2012. Αλλά θα ήθελα να σας ε, ερωτήσω τι, για ποιο λόγο τέσσερις χώρες είχαν την ευθύνη για 16% όλων των δημοσιονομικών 60% συγγνώμη, όλων των δημοσιονομικών διορθώσεων που επήλθαν το 12. Αυτό είναι κάτι το οποίο φαίνεται παράδοξο σε σχέση με την ε, λειτουργία του προϋπολογισμού όταν 20 κράτη-μέλη έχουν λειτουργήσει θετικά και τα ασφάλματα τα οποία βλέπουμε για, την, ε, για τον προϋπολογισμό εστιάζονται πάντα στα ίδια κράτη. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα λοιπόν. Γιατί συμβαίνει αυτό. Το δεύτερο έχει να κάνει με το Ελεκτικό συνέδριο. Λέει το Ελεκτικό συνέδριο ότι εδώ και πολλά χρόνια τα ίδια τα κράτη-μέλη αυτά θα έπρεπε να είχαν διαπιστώσει όλα αυτά τα σφάλματα τα οποία ανεκάλυψε στη συνέχεια το ε, ελεκτικό συνέδριο τα οποία σε ορισμένε περιπτώσεις ήταν πολύ μεγάλο ποσοστό σφαλμάτων. Πώς λοιπόν μπορούμε εμείς να αντιμετωπίσουμε αυτό το έργο του ελέγχου και να το αφήνουμε απόλυτα στο έργο των εθνικών κρατών. Φυσικά δειγματοληπτικά το ελεκτικό συνέδριο κάνει ελέγχους και διαπιστώνει ότι τα σφάλματα αυτά τα οποία ανεκάλυψε θα έπρεπε να είχαν ήδη ανακαλυφθεί μέσα στα ίδια τα κρατημέλη. Με ενδιαφέρει λοιπόν να μπορέσουμε να έχουμε ένα αξιόπιστο σύστημα ε, ελέγχου, αλλά αυτό εξαρτάται και από το έργο των εθνικών ελεκτών. Θέλω πλέον να πω ότι για κατά 90% λειτουργεί πολύ καλά το σύστημα της διαμεμοιρασμένης διαδικασίας εκτέλεσης του προϋπολογισμού όπως στον τομέα της υγειοργίας και τα λοιπά. Αλλά αναρωτιέμαι πώς μπορείτε εσείς να καταλήγετε στο συμπέρασμα ότι εμείς ως ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωρίζοντας το επίπεδο των ε, σφαλμάτων να δώσουμε απαλλαγή για το έτος 2012. Ένα τρίτο ερώτημα που θέλω να θέσω έχει να κάνει με το θέμα της αναγνώρισης και του ελέγχου της έκτασης των αγροτεμαχίων. Το ελεκτικό συνέδριο σε 21 κράτη τα τελευταία χρόνια έχει διαπιστώσει την ύπαρξη προβλημάτων. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάλι εκφράζει επιφυλάξεις για τρία κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του συστήματος αυτού. Θεωρεί το σύστημα αυτό δεν λειτουργεί ικανοποιητικά και δεν μπορεί επομένω να εκτιμήσει αν θα βελτιωθούν όλα αυτά τα πράγματα στο άμεσο μέλλον. Θα ήθελα να ξέρω πώς δεδομένων όλων αυτών, όταν η ίδια η Κομισιόν εκφράζει επιφυλάξεις για τα ζητήματα αυτά, πώς εσείς μας ζητάτε να δώσουμε την απαλλαγή σε αυτή την περίπτωση. Και θα ήθελα να θέσω και ένα ερώτημα ειδικά για την Ελλάδα πώς ε, βλέπετε το σύστημα αυτό να λειτουργεί με τις δημοσιονομικές διορθώσεις για το σύστημα ελέγχου των επιδοτήσεων των εκτατικών και φαίνεται ότι κατά κάποιο, σε κάποιο βαθμό δεν ήταν επακριβείς οι πληροφορίες και οι αιτήσει που έγιναν για τις επιδοτήσεις αυτές. Ένα ακόμα ερώτημα για την αγροτική ανάπτυξη. Δυστυχώς εδώ βρίσκεται το υψηλότερο ποσοστό σφαλμάτων και εσείς ο ίδιος Είπατε ότι οι διορθώσεις οι οποίες προβλέπονται για το νέο αυτό σύστημα θα λειτουργήσουν μόνο ε, σε μερικά χρόνια, σε, του, του χρόνου μάλλον. Αλλά μας λέτε παρόλα αυτά ότι πρέπει να δώσουμε την απαλλαγή. Σε τι βασίζεται την προσδοκία σας ότι στο άμεσο μέλλον θα υπάρξει δυνατότητα το σύστημα αυτό να λειτουργήσει ορθά. Και μια τελευταία παρατήρηση για την ε, περιφερειακή πολιτική. Εδώ το, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 16 κατημέρες ό,τι αφορά το περιφερεια, τα περιφερειακά ταμεία και την, ε, ε, το Μείο Συνοχής έχει εκφράσει τις επιφυλάξεις της. Και πάλι πρέπει να σας θέσω το ερώτημα ως, εκπροσώπου του, ως εσάς ως εκπρόσωπο του Συμβουλίου γιατί προτείνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει την απαλλαγή παρά αυτά τα σχόλια της Κομισιόν. Ευχαριστώ τον εισηγητή μας κύριο Πίπερ και να ανοίξω τώρα τη συζήτηση. καλό τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων, πρώτος ο κύριος Γκάιερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, και εγώ σας καλωσορίζω στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Υπουργέ που είστε εδώ ενώπιόν μας για να μας παρουσιάσετε την άποψη του Συμβουλίου των Υπουργών και χαίρομαι ιδιαίτερα για την ανάλυση που περιέχει η έκθεση γιατί πρώτη φορά βλέπω να αναφέρεται σε ένα έγγραφο του Συμβουλίου τόσο αναλυτικά ο ρόλος των κρατών μελών και σε πολλά σημεία αναφέρεστε στα προβλήματα που έχουν τα κράτη-μέλη για να ε, διαχειριστούν και να ελέγξουν τον τρόπο ε, δαπάνησης των ε, ενωσιακών πόρων. Ακόμη και το έγγραφο των τριών Υπουργών Οικονομικών που είναι κατά της απαλλαγής αναφέρουν πολύ σαφώς τον ρόλο των κρατών μελών είναι πολύ σαφή αυτά. Βεβαίως ο συνάδελφος Δόκτωρ Πίπερ αιτιολογημένα επικρίνει τα συστήματα ελέγχου των κρατών μελών. Το ερώτημά μου είναι τι συμπεράσματα εξάγεται από αυτή την ανάλυση. Και νομίζω ότι μόνο δύο συμπεράσματα μπορεί να εξάγει κανείς. Πρώτον, είτε το Συμβούλιο θα έπρεπε να δώσει συνέχεια στην άποψή του, το οποίο κατά τη γνώμη μου θα σήμαινε απλά και μόνο ότι θα έπρεπε να γίνει μια αποτίμηση από ομότιμους των αποτελεσμάτων. Δηλαδή, θα έπρεπε να αρχίσουν να συζητούν μεταξύ τους Υπουργοί Οικονομικών, για το τι πρέπει να βελτιώσει ο καθένας στον τομέα αρμοδιότητάς του Ε, να κλείσω τώρα τη συζήτηση για το θέμα αυτό, γιατί αλλιώ θα μπω σε ε, τομεί πολιτική φαντασία. Αλλά αυτή θα ήταν μία δυνατή επίπτωση. Και το άλλο θα ήταν να επιτρέψουμε στην Κομισιόν να ελέγχει εντονότερα τα συστήματα διαχείριση στα κράτη-μέλη. Δηλαδή, ω Επιτροπή Ελέγχου του Υπροπολογισμού, μαζί με το Συμβούλιο, συμφωνούμε για του στόχου που πρέπει να θέτουμε για τη δαπάνη των πόρων. Συμφωνούμε ότι τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων των 28 κρατών μελών πρέπει να αξιοποιούνται για να επιτυχάνουμε πολιτικούς στόχους με καλύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο και με τρόπο και πιο διαφανή προς τους ε, ψηφοφόρους. Αλλά πώς θα το επιτύχουμε. Το Συμβούλιο ξεκινά μια συζήτηση για το ρόλο των κρατών μελών. Αυτό νομίζω ότι είναι πραγματική πρόοδος. Αυτός είναι ο τρόπος για να πάμε ακόμη καλύτερα. Ο Επίτροπος Εμέτα, στη σύντομη δήλωσή του, είπε, και σε αυτό συμφωνεί η Επιτροπή μας, και μας το είπε και ο πρόεδρος του Λεγκτικού Συνεδρίου, όταν μας παρουσίασε την ετήσια έκθεση του, πόσα λάθη θα έπρεπε να έχουν ήδη διαπιστωθεί στα κράτη-μέλη. Υπάρχουν λοιπόν πολλές δυνατότητες ε, που θα μπορούσε να αξιοποιήσει το Συμβούλιο, να υπάρξει δηλαδή ένας ε, θεσμικός διάλογος. Θα ήταν ε, κάτι το πολύ θετικό. Εάν λοιπόν θέλουμε να διερευνήσουμε περαιτέρω πώς μπορούν τα κράτη-μέλη να αξιοποιήσουν καλύτερα τους ενωσιακούς πόρους, νομίζω ότι θα οδεύαμε προς σωστή κατεύθυνση και επαναλαμβάνω ότι χαίρομαι για την παρουσία και την παρουσίαση σας κύριε ε, Υπουργέ. Ο κύριος Γκόραν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ χαιρετίζω την παρουσία του Υπουργού αλλά και του Επιτρόπου ο οποίος τόνισε ιδιαίτερα την ευθύνη των χωρών μελών ενώ ο υπουργό της Κομισιόν. Κατανοητό, γιατί εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε πάντα στη μέση των, μεταξύ των δύο και προσπαθούμε να ζυγιάσουμε ποιος φταίει. Τα τρία κράτη-μέλη που δεν ενέκριναν την απαλλαγή νομίζω ότι το θέμα εδώ δεν είναι καθόλου απαλλαγή, <clears throat> είναι καθαρά πολιτικό για πολιτικούς λόγους την απέρριψαν και δεν ε, ήταν θέμα καθαρά λογιστικό. Τώρα αν δούμε τους αριθμούς η Κομισιόν έχει κάποιο δίκιο αλλά και εμείς όταν λέμε ότι 80% της χρήσης του προπολογισμού είναι ευθύνη των χωρών μελών όταν λέει η Κομισιόν μάλλον άρα φέρουν και το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης έχει κάποια λογική αυτό και πολλοί από εμά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα θέλαμε στο μέλλον τα κράτη-μέλη που θεωρούνται προβληματικά, γιατί τα μικρότερα κράτη είναι τα πιο προβληματικά, να ψεχθούν και αυτά δεόντως. Τώρα για το Συμβούλιο συγκεκριμένα. Θεωρείται ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στη συμπεριφορά ορισμένων χωρών μελών, παραδείγματος χάρη ένα σχέδιο δράσης από την Κομισιόν για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που δημιουργούν οι πιο προβληματικές αυτές χώρες μέλη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζούμπιχ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ τον ε, Υπουργό και τον Επίτροπο γιατί όλοι επιθυμούμε να αξιολογήσουμε αντικειμενικά τη δραστηριότητα των κρατών μελών και χαίρομαι που υπάρχει διαφάνεια για το ποστό σφαλμάτων. Για όλους μας είναι θετικό αυτό, ότι γίνονται σωστοί έλεγχοι και όταν υπάρχουν σφάλματα να αναφέρονται δημοσίως και να συζητιώνται και εδώ στην Επιτροπή μας ζωντανά στο διαδίκτυο επίσης. Αυτό αποδεικνύει ότι όλοι κάνουμε κάθε προσπάθεια να μειωθούν στο μέλλον τα σφάλματα αυτά. Αλλά το ερώτημα είναι τι βήματα θα αναλάβουμε ούτω ώστε στα κράτη-μέλη που υπάρχουν πολλά σφάλματα να βελτιωθεί η κατάσταση. Μία κεντρική απέτηση είναι αυτή. Και επίσης ε, θα πρέπει να καταρτήσουμε τους αρμοδίους. Να έχουν καλύτερη κατάρτιση λοιπόν για να βελτιωθεί η κατάσταση. Ερώτημα από πλευρά μου. Υπάρχουν βέλτιστες πρακτικές, υπάρχουν κριτήρια αξιολόγηση, υπάρχουν στατιστικές πώς ε, ε, βοηθάμε και πώς επιμορφώνουμε τους αρμόδιους στις διάφορες εθνικές υπηρεσίες. Υπάρχουν γενικότερα αντιλήψεις πώς μπορούμε να βοηθήσουμε μέσω αγωγής τεχνολογίας, ε, πώς μπορούμε να τους κάνουμε μαθήματα. Ξέρουμε ότι υπάρχει δυνατότητα e-learning, ηλεκτρονική εκμάθηση. Μπορεί να βοηθήσει. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να εισαγάγουμε το ISO 9000 ούτως ώστε να έχουμε καλύτερες διαδικασίες διότι βεβαίως εάν χορηγήσουμε επιμόρφωση εάν δώσουμε βοήθεια οπωσδήποτε θα μειωθεί κατά πολύ το ποσοστό σφαλμάτων έχει η Κομισιόν προτάσει για το θέμα αυτό και το Συμβούλιο έχει πρόθεση να βοηθήσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω κάποιον άλλο μιλτή από τα μέλη της Επιτροπής μας και θα ήθελα να σας δώσω και πάλι το λόγο κύριε Υπουργέ για να απαντήσετε. Ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας, για τις ε, κριτικές σας παρατήρησεις και τα ερωτήματά σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω ε, τα ερωτήματα αυτά όσο μπορώ στο σύντομο χρόνο που έχω στη διάθεσή μου. Ένα γενικό σχόλιο πρώτα. Όλοι μας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Κομισιόν και το Συμβούλιο, συμμεριζόμαστε τις ίδιες αξίες και έχουμε τους ίδιους στόχους. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε αποτελεσματική προστασία του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια ε, αποτελεσματική και ε, ορθή διαχείριση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την σωστή εφαρμογή των κανόνων για να υπάρξει πλήρη συμμόρφωση από όλους. Νομίζω ότι πρέπει να συνεργαστούμε σε αυτό το κοινό έδαφος για να είμαστε αποδοτικοί και αποτελεσματικοί και να εξασφαλίσουμε ότι τα προγράμματα και τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίδουν τα σωστά αποτελέσματα με ένα σαφή και ορθό τρόπο. Αναφερθήκατε στις τέσσερις χώρες τις τρεις χώρες που δεν υποστήριξαν τα, τη σύσταση του Συμβουλίου. Αλλά 25 χώρες, οι υπόλοιπες χώρες, δεχτήκανε αυτή τη θέση. Τα τρία κράτη-μέλη ανέφεραν ε, ότι γνωρίζουν, αναγνώρισαν τα αποτελέσματα του ελεκτικού συνεδρίου, αλλά θα θέλανε να υπάρξει περισσότερη ε, βελτίωση στην ε, οικονομική διαχείριση, δημοσιονομική διαχείριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2012 σε σχέση με τον προϋπολογισμό. Τονίζουν ότι είναι έτοιμοι να αναλάβουν την πλήρη ευθύνη του να εφαρμόσουν πλήρες και αποτελεσματικούς κανόνες για τη διαχείριση των ποσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζήτησαν να υπάρξουν περαιτέρω μέτρα τα οποία θα ληφθούν για καλύτερα αποτελέσματα. Πιστεύω τώρα ότι ήδη και στην ομιλία μου <clears throat> συμπεριέλαβα ορισμένες από αυτές τις ε, επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν και τις προτάσεις και υπάρχει ένα κοινό έδαφο υποστήριξης για μια πιο αποτελεσματική και διάφανη χρήση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, για το θέμα που ετέθη σε σχέση με τη θέση του Συμβουλίου. Είναι σημαντικό το θέμα αυτό που αναφέρατε. Το Συμβούλιο έχει καταγράψει την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως έχει εκφραστεί σε διάφορα ψηφίσματα ολομελίας θέλω να καταστήσω σαφές και αυτό είναι ένα γενικό πολιτικό θέμα ότι το Συμβούλιο συμφωνεί ότι όλες οι δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι διοικητικές δαπάνες φυσικά πρέπει να τη χάνουν προσεκτικού ελέγχου από τους αρμόδιους φορείς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την απόδοση της απαλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο πρέπει να είναι σε θέση να διερευνήσουν την ε, αποτελεσματικότητα και την ποιότητα της, του δημοσιονομικού, δημοσιονομικής διαχείρισης των ε, άλλων οργάνων, το κάθε όργανο για το, για τον, ε, για το, το Συμβούλιο για το Κοινοβούλιο και τούμπαλιν. Μας ενδιαφέρει να διεδρεώσουμε μακροπρόθεσμα, σε μακροπρόθεσμο επίπεδο ένα σύστημα συνεργασίας για να μπορούμε να βρίσκουμε κοινό έδαφος σε επίπεδο ισότητος. Έχει προταθεί να υπάρξει μια Συμφωνίασε στο θέμα αυτό. Αυτή η πρόταση έχει ήδη διατυπωθεί το Σεπτέμβριο του 2010 για ένα μνημόνιο κατανόησης το οποίο θα καλύπτει τη διαδικασία αμοιβαία χορήγησης απαλλαγή. Κάτι που διατυπώθηκε ω πρόταση το 2011. Συμφωνή, θεωρεί το Συμβούλιο ότι είναι σημαντικό να μπορέσουμε να βρούμε μια συμφωνία για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, ώστε να εξασφαλιστεί η αμοιβαία λογοδοσία και διαφάνεια με πλήρη σεβασμό βέβαια των αρμοδιοτήτων κάθε θεσμικού οργάνου βάσει της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατανοώ από τις πρόσφατες άτυπες επαφές που έγιναν μεταξύ Προεδρίας και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι ο δικός σας θεσμός θα ήθελε να ε, προωθήσει περαιτέρω το διάλογο αυτό με το Συμβούλιο σε σχέση με το θέμα της απαλλαγής του Συμβουλίου. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι το Συμβούλιο είναι έτοιμο να προχωρήσει σε συζητήσεις με στόχο να υπάρξει συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ταχύτερο δυνατό. Για τις εθνικές δηλώσεις που αναφέρθηκε προηγουμένως. Ξέρετε ότι είναι ένα πολύπλοκο θέμα με πολλές διαστάσεις που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη με τον νέο δημοσιονομικό κανονισμό ιδιαίτερα που έχει τεθεί σε εφαρμογή από το 2013 έχουν επέλθει αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η λειτουργία του προεπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με επιμερισμένη διαχείριση. Μεταξύ άλλων υπάρχει η πρόνοια ότι τα, οι φορεί των κρατών μελών που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των κονδυλίων αυτών θα δίδουν μια δήλωση διαχείρισης στην Κομισιόν σε σχέση με το έργο τους. Και επίσης σε εθελοντική βάση τα κάτι μέλη μπορεί να δώσουν εθνικές δηλώσεις εφόσον το επιθυμούν και οι οποίες θα πρέπει να προερχόνται από το αρμόδιο επίπεδο. Η συμβαστική λύση που έχει προβλεφθεί για τον κανονισμό αυτό, το νέο δημοσιονομικό κανονισμό, είναι το αποτέλεσμα μακρών και δυσκόλων διαπραγματεύσεων, κατά την άποψη του Συμβουλίου. Αυτή η συμβαστική λύση για το δημοσιονομικό κανονισμό έχει εξεύρει τη σωστή ισορροπία μεταξύ της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το θέμα αυτό. Συγχρόνως, το Συμφούλιο συμφώνησε να συμμετάσχει στο έργο της διαθεσμικής ομάδος εργασίας για τις εθνικές, για τις εθνικές δηλώσεις που ξεκίνησε το 2013 με πρωτοβουλία της Κομισιόν ετήσι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ομάδα αυτή δεν έχει συμπληρώσει το έργο της σε σχέση με τις συστάσεις οι οποίες θα πρέπει να διατυπωθούν και συνεχίζει την επεξεργασία της. Να σας υπενθυμίσω ότι οι συστάσεις αυτές δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα και δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε όλα τα κράτη-μέλη με ε, ε, ενιαίο τρόπο. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι θα πριτανεύσει μια επικοδομητική αντιμετώπιση μέσα σε αυτή την ομάδα η οποία θα μπορέσει να συμπληρώσει το έργο της σύντομα. Πιστεύω ότι οι διαδικασίες λογοδοσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ενισχυθούν για να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια στον, στην εκτέλεση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Η ανάγκη όμως να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να είναι αντικείμενο βαθιάς ε, συζήτησης και διαβούλευσης. Περιμένουμε, πρέπει να περιμένουμε λοιπόν τις συστάσεις αυτής της ομάδας εργασίας. Για τις δημοσιονομικές διορθώσεις και τις ανακτήσεις που αναφέρατε προηγουμένως. Όπως είπα προηγουμένως, είναι κέρυες αυτές οι ανακτήσεις και διορθώσεις για να προστατευτεί ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Συμβούλιο μπορεί να επιβεβαιώσει και πάλι την Κομισιόν για τη συνέχιση τη εφαρμογή δημοσιονομικών διορθώσεων και ε, ανακτήσεων, ιδίως σε ό,τι αφορά τις μη κανονικά δαπανηθήσει ε, πιστώσεις. Μας ενδιαφέρει να ενισχύσουμε τα ελεκτικά συστήματα, να συνεχίσουν προσπάθειες στον τομέα αυτό και να εφαρμοστεί μια σαφής πολιτική για την αναστολή ή τη διακοπή πληρωμών όταν υπάρχει αποχρόν λόγος. Αυτό αφορά φυσικά και την Ελλάδα, γιατί με ρωτήσατε για τη δική μου χώρα και εφόσον θέσατε αυτό το ερώτημα, θέλω να κάνω κάποια σχόλια. Οι ελεγκτές για τη χώρα μου είχαν κάποια ε, πορίσματα στην έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου για το 2012 σε ό,τι αφορά διαρθωτικά θέματα στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης και της πολιτικής συνοχής. Παρ' όλα αυτά, τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε σημαντική πρόοδος σε ό,τι αφορά το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης και ελέγχου στην Ελλάδα. Και ιδιαίτερα η πρόοδος αυτή έχει επιτευχθεί στους κατωτέρω τομείς. Εντατικοποίηση των ελέγχων από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, ενίσχυση της στρατηγικής ελέγχου και εντατικοποίηση των διαδικασιών, βελτίωση της ποιότητας των υποβαλωμένων προτάσεων από δυνητικούς δικαιούχους, που είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση χάρη στο καλύτερο σύστημα ελέγχου, πιο αποτελεσματική επίτευξη του σχεδίου για ε, πολλαπλή συμμόρφωση επί τη βάση των προτάσεων της Κομισιόν. Όλα αυτά έχουν βελτίωσει το, έχουν μειώσει το επίπεδο σφαλμάτων το χρονικό διάστημα 2012-2013, όπως αναφέραν οι εθνικές ελεγκτικές αρχές το ποσοστό αυτών σφαλμάτων. Την περίοδο 2012-2013 μειώθηκε στα 2, έφτασε το 2,6% από 4,9% που ήταν την προηγούμενη περίοδο 2011-2012. Προς την κατεύθυνση αυτή επίσης, η, ο Υπουργό Οικονομικών της χώρας μου συνεχίζει τις προσπάθειες βελτίωσης, εστιάζοντας τον καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών ε, πάταξη της απάτης, την ενίσχυση της λειτουργικής ικανότητας των αρμοδίων υπηρεσιών, την, ε, το σχεδιασμό για την καταπολέμηση της απάτης το 2014 και την περαιτέρω βελτίωση των διαδικασιών ελέγχου για τα αγροτικά θέματα και την ανάπτυξη. Βεβαίως, το Συμβούλιο έχει εκφράσει την απογοήτευσή του ε, για τα σφάλματα αυτά, για την αύξησή τους μάλιστα. Ωστόσο, Πρέπει να ε, ε, διαπιστώσουμε ποια είναι τα προβλήματα ακριβώς. Και το συνέδριο τα διαπίστωσε ότι δεν ε, γίνονται σεβαστά τα κριτήρια ευλεξιμότητας δηλαδή γίνεται υπερβολική δήλωση επιφανειών, δεν γίνονται σεβαστές οι αγροπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις και δια παράβαση άλλων κανόνων, αλλά βέβαια τα προγράμματα αυτά είναι πολύ περίπλοκα. Το Συμβούλιο συμφωνεί πλήρως με τις δράσεις που προτείνει να αναλάβει η Κομισιόν και καλεί την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν ε, σύντομα τα προγράμματα δράση που έχουν ε, διατυπωθεί και όλα τα αναγκαία προληπτικά διορθωτικά μέτρα. Και η Επιτροπή ήδη έχει εφαρμόσει ορισμένα αυτά τα μέτρα. Για παράδειγμα, στη Γεωργία η Επιτροπή ε, έχει προχωρήσει στη διαδικασία εκαθάρισης των λογαριασμών και όπου είναι αναγκαίο έχει διατυπωθεί και πρόγραμμα δράση. Τα τελευταία πέντε χρόνια τα προγράμματα δράση έχουν αρχίσει να λειτουργούν σε πέντε κράτη-μέλη. Στον τομέα τη ανάπτυξη τη υπαίθρου, του περιβάλλοντο, τη αλληλεία και τη υγεία. Το 2012 ε, ε, εκπονήθηκαν για 14 κράτη-μέλη το 12 και θα επεκταθούν σε όλα τα κράτη-μέλη το 2013. Η Επιτροπή επίσης μας ενημέρωσε ότι διάφορα κράτη-μέλη τροποποίησαν τα προγράμματά τους ανάπτυξης της υπαίθρου για να διευκρινιστεί ή για να αλλάξει η κατάσταση όσον αφορά τους, ε, τις συνθήκες για ενωσιακή χρηματοδότηση. Τέλος, επαναλαμβάνω να σας για άλλη μια φορά ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων. Με χαρά ε, διαπίστωσε ότι ε, συμμεριζόμεθα πολλές ανησυχίες και επίσης ε, ότι είναι μέλημά μας να υπάρξει πρόοδος κάθε χρόνο για να δημιουργηθεί η βάση για μια ανεπιφύλακτη θετική γνώμη του συνεδρίου. Καλώ όλους τους εμπλεκόμενους, Κοινοβούλιο, Επιτροπή, Συμβούλιο, το Συνέδριο και τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν επικοδομητικά για να επιτευχθεί χρηστή οικονομική διαχείριση και έλεγχος της ενωσιακής χρήσης πόρων. Είναι σημαντικότερο σήμερα παρά ποτέ να δείξουμε την δέσμευσή μας και να καλέσουμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να αναλάβουν πλήρως τις ευθύνες τους και να ασκήσουν προσεκτικά τον ελεγκτικό και επιτηρητικό τους ρόλο. Πρέπει να υπάρξει περαιτέρω. Πρόοδος τα επόμενα χρόνια. Πρέπει να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα προς τους Ευρωπαίους πολίτες και φορολογούμενους ότι οι ενωσιακοί πόροι χρησιμοποιούνται με υπεύθυνο και διαφανή τρόπο. Πιστεύουμε ότι η νέα πολιετής περίοδος προγραμματισμού είναι μια σημαντική ευκαιρία να υπάρξει μεγάλη πρόοδος προς την απλούστευση και άρα τη μείωση του κινδύνου σφαλμάτων αξιοποιώντας τεχνολογικές δυνατότητες όπως αναφέρθηκε. Είναι μια ευκαιρία για στενή συνεργασία των θεσμικών οργάνων της Ένωσης ούτως ώστε να εκπονήσουμε νέες πρωτοβουλίες για να εμπλουτίσουμε και το πλαίσιο και τις διαδικασίες που αφορούν την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Τέλος, να κάνω ένα σχόλιο στα ελληνικά, γιατί θίξατε μερικά θέματα. Ε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και μέλη της Επιτροπής για τα πολύ θετικά του σχόλια που κατέθεσαν για την τεράστια προσπάθεια που καταβάλει η ελληνική κυβέρνηση και οι Έλληνες πολίτες. Με τη βοήθεια τη δική σας, με τη βοήθεια των εταίρων. Η Ελλάδα πλέον πετυχαίνει και οι αριθμοί το επιβεβαιώνουν το 2013 να αντιμετωπίσει τα υψηλά διαχρονικά δίδυμα ελλείμματά της. Θα επιτύχει το 2013 σημαντικό πρωτογενές πλεόνασμα και ήδη επέτυχε πλεόνασμα στο συζύγιο των συναλλαγών μετά από πάρα πολλές δεκαετίες. Άρα η χώρα οδεύει προς την έξοδο από την κρίση. Και προς την κατεύθυνση αυτή θα συνεχίσουμε ώστε να πιάσουν τόπο οι τεράστιες θυσίες των Ελλήνων πολιτών και η αρρωγή αλλά και η αλληλεγγύη η δική σας των εταίρων. Ladies and gentlemen, honorable members of the ε, Κυρίε και κύριοι, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σα εύχομαι ό,τι καλύτερο για την εργασία σα τι επόμενε εβδομάδε στα πλαίσια τη διαδικασία απαλλαγή για το 2012. Ευχαριστώ πολύ. Thank Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Υπουργέ, για τις δηλώσεις σας και τις απαντήσεις σας χαιρόμαστε ιδιαίτερα που μας ανακοινώσατε το Συμβούλιο είναι διατεθειμένο να αναζητήσει μια λύση για το πρόβλημα της απαλλαγής και να υπάρξει επιτέλους κάποια πρόοδο σε αυτό το πολύ ζωτικό θέμα. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ξέρουμε ότι είναι πολύ βεβαρημένο το πρόγραμμα πάντοτε των προεδρευόντων και Γι' αυτό εξ ονόματος όλη μας της Επιτροπής εύχομαι στην Ελληνική Προεδρία καλή επιτυχία γιατί όλοι χρειαζόμαστε επιτυχίες για, να, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά τις επικρίσεις που είναι και αυτές απαραίτητε. θέλουμε όλοι να βελτιωθούν τα αποτελέσματα και να υπάρξει πρόοδος. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ για την παρουσία σας και καλή τύχη ιδιαίτερα για τις εξελίξεις στην Ελλάδα που είναι και προς το συμφέρον του λαού όπως είπατε και εσείς. Ευχαριστώ. <laughs> <laughs>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 Αγαπητοί συνάδελφοι, μετά από την ε, παρουσίαση της ελληνικής προεδρίας από τον κύριο Σταϊκούρα, θα ήθελα τώρα να υποδεχτώ μια εκπρόσωπο της Ισπανικής κυβέρνησης, την ε, Υφυπουργό για θέματα προϋπολογισμού και δημοσίων δαπανών του Ισπανικού Βασιλείου, κυρία Φερνάντες Κουράς. Καλώς κυρία Κουράς. Στην Επιτροπή μας πρόκειται για μια πρωτοβουλία του κυρίου Πίπερ, ο οποίος σας κάλεσε, ώστε να μπορέσετε στη διαδικασία, στα πλαίσια της διαδικασίας απαλλαγής να λάβετε το λόγο ενώπιον της ε, Επιτροπής μας και θα ήθελα να δώσω και πάλι το λόγο στον ε, εισηγητή, τον κύριο Μάρκους Πίπερ, ο οποίος είχε ένα συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο ήθελε να σας προσκαλέσει εδώ και να έχουμε τη δυνατότητα βελτίωσης του δημοσιονομικού ελέγχου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλώς ήρθατε, Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας κύριε Πίπερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήλθατε κυρία Κουράς, κυρία Υφυπουργέ. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την παρουσία σας και για το γεγονός ότι μπορούμε να αναφερθούμε στην ιδιαίτερη κατάσταση στην Ισπανία. Η Ισπανία όπως ξέρουμε είναι ένα ομοσπονδιακό κράτος όπως και η Γερμανία. Στη Γερμανία έχουμε αντιμετωπίσει και εκεί σημαντικά προβλήματα για την ε, εφαρμογή των κονδυλίων του Κοινωνικού Ταμείου και στην δική μου περιοχή, την Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία, υπήρξε σε κάποια στιγμή αναστολή της χορήγησης πιστώσεων, κάτι το οποίο είναι γνωστό. Θα ήθελα εδώ να αναφερθώ στην κατάσταση η οποία ισχύει στην Ισπανία γιατί τα τελευταία χρόνια υπήρξαν βελτιώσεις. Φαίνεται ότι λειτουργεί η νέα πολιτική η οποία εφαρμόστηκε. Από την άλλη πλευρά εξακολουθεί να υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο προβλημάτων. Για το 2012 από τα 13 δισεκατομμύρια που πήρε συνολικά η Ισπανία στην επιμερισμένη διαχείριση υπήρξαν διορθώσεις του ύψους του 2,1 16,8 του συνόλου. Αυτό είναι ένα υψηλό επίπεδο. Ενδεχομένως θα, μπορείτε να μας, θα μπορούσατε να μας πείτε τι έγινε στην περίπτωση αυτή και όλα αυτά τα σφάλματα τα οποία παρουσιάστηκαν στην περίοδο 2000-2006 δεν μπόρεσε να διορθωθούν και είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε διορθώσεις το 2012. Αυτό είναι κάτι το οποίο οδηγεί σε ουσιαστικά προβλήματα στη χρησιμοποίηση των κονδυλίων. Το 2012 η Κομισιόν μας είπε ότι για 23 προγράμματα στην Ισπανία εκφράζει επιφυλάξεις. Αυτή είναι μια κατάσταση που εγώ δεν μπορώ να δεχθώ ως φυσιολογική και δεν μπορώ να την κρίνω, αλλά ίσως θα μπορούσατε εσείς από τη δική σας ε, την ισπανική οπτική γωνία να μας εξηγήσετε γιατί προέκυψαν αυτές οι επιφυλάξεις που αν, είχε, αν ήταν με θέματα εποπτείας τα προβλήματα, που βρεθήκαν οι δυσκολίες οι οποίες προέκυψαν και αν θα μπορούσατε να δώσετε μια απάντηση η οποία θα ε, ενημερώσει καλύτερα και θα διαφωτίσει την Επιτροπή μας. Έχουμε ακούσει από το Ελεκτικό Συνέδριο εδώ και πολλά χρόνια, συνεχίζεται αυτό, ότι περίπου 60% των σφαλμάτων ε, είναι σφάλματα τα οποία θα έπρεπε να είχαν αποκαλυφθεί από τα ίδια τα κράτη-μέλη. Και έχουμε ένα σύστημα ελεκτικό το οποίο βασίζεται στην ορθή λειτουργία του ελέγχου και στα κράτη-μέλη. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο ίσως θα θέλατε να αναφερθείτε σε λεπτομεριακό επίπεδο περισσότερο για την κατάσταση της Ισπανίας, πώς μπορεί κανείς να επανορθώσει τις δυσκολίες και τα σφάλματα αυτά και πού θα μπορούσε να παίξει κάποιο ρόλο να σας βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά είναι τα ερωτήματα που ήθελα να σας θέσω. Ευχαριστώ τον εισηγητή, τον κύριο Πίπερ για τις εισαγωγικές του παρατηρήσεις και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Μάρτα Φερνάντες Κουράς και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας σε όλους και όλες. Είμαι ενώπιον σας σήμερα ως Υφυπουργός Οικονομικών για τα θέματα προϋπολογισμού και δημοσίων δαπανών. Είμαι αρμόδια για τα θέματα των Περιφερειακών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής και είμαι επικεφαλής διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων στην Ισπανία. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να εκφράσω την ικανοποίησή μου και τις ευχαριστίες μου στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που μου έδωσε την ευκαιρία να παρουσιάσω και το επίπεδο της διαχείρισης των κονδυλίων αυτών στην Ισπανία, αλλά και το παρελθόν και το προσδοκόμενο μέλλον για τα κονδύλια αυτά. Ένα θέμα μεγάλη σημασία σχετικά με όλα αυτά. Είναι ένα θέμα μάλλον πολύ σημαντικό αυτό για τη χώρα μας, γιατί ήμασταν από τους κυριότερους αποδέκτες κονδυλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστεύω ότι μπορέσαμε να εκμεταλλευτούμε πάρα πολύ θετικά αυτά τα κονδύλια, όπως διαπιστώνουν όλοι αυτοί οι οποίοι ταξιδεύουν στην Ισπανία, όπως εσείς ή όλοι αυτοί που έχουν παρακολουθήσει την εξέλιξη των οικονομικών δικτών στη χώρα μας. Παρ' όλα αυτά, τα αποτελέσματα αυτά που επετέθησαν με τη βοήθεια ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι αυτό στο οποίο θέλω να σταθώ. Θέλω να σταθώ σε ένα άλλο σημείο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, που είναι η σωστή διαχείριση και ο έλεγχος των κονδυλίων σε όλη αυτή την μακρόχρονη διαδικασία και μιλώ για μια διαδικασία ή καλύτερα για ένα δρόμο, μια πορεία που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς πόρους. Από τότε που η Ισπανία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αλλάξει σημαντικά η φύση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά, όλες αυτές οι αλλαγές μας έχουν υποχρεώσει να προβούμε σε μια βαθμία προσαρμογή και να δείξουμε ευκαμψία και ικανότητα αντίδρασης. Και φυσικά με τον τρόπο αυτό, αυτά τα θέματα οδήγησαν σε αντιμετώπιση ιδιαίτερων προβλημάτων στην Ισπανία που θέλω να τονίσω. Πολλοί εκπλήσονται για το γεγονός ότι η Κομισιόν στην έκθεση της του 2012 αναφέρει ότι στην περίοδο προγραμματισμού 2000-2006 η Κομισιόν προέβη Ε, σε δημοσιονομικές διορθώσεις 2,26 ε, δισεκατομμυρίων ευρώ, που είναι περίπου το 16% του συνόλου. Επίσης, πολλοί εκπλήσονται για το γεγονός ότι το ελεκτικό συνέδριο σε σχέση με το οικονομικό έτος 2012 σε ό,τι αφορά την Ισπανία αναφέρει σαν παράδειγμα διαδικασίας διανομικής διόρθωσης το ίδιο αυτό ε, αντικείμενο που έχει να κάνει με 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ σε ό,τι αφορά την εφαρμογή κονδυλίων συνοχής στο χρονικό διάστημα 2000-2006, γιατί είναι η μεγαλύτερη μεμονωμένη ε, διόρθωση του 2012 ε, με ποσοστό 49%. Για να μπορέσουμε να καταλήξουμε λοιπόν καλύτερα το περιεχόμενο της έκθεσης Κομισιών και του Ελεκτικού Συνεδρίου για το θέμα αυτό, θέλω να κάνω κάποιες διευκρινήσεις. Πρέπει να κάνω κάποιες διευκρινήσεις. Πρώτα απ' όλα θέλω να αναφέρω ότι οι οικονομικές αυτές διορθώσεις που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς της Κομισιόν το 2012 έχουν να κάνουν με δαπάνες που έχουν γίνει με προληπτικό τρόπο από τις Ισπανικές Αρχές και επομένως με πρωτοβουλία Ισπανική για το χρονικό διάστημα 2006 και πριν από το τέλος του 2010 όταν σταμάτησαν τα λειτουργικά αυτά προγράμματα του χρονικού διαστήματος 2000-2006 έγιναν αυτές οι ενέργειες. Δεν είναι κάτι που αναδύεται λοιπόν ξαφνικά το 2012. Είναι κάτι το οποίο οφείλεται σε αλλαγή μεθοδολογίας ό,τι αφορά την παρουσίαση των στοιχείων από την Κομισιόν. Το γνωρίζει και η Κομισιόν και το αναγνωρίζει στα σχόλιά της στο παράρτημα 1 του, της έκθεσης του ελεκτικού συνεδρίου, η, ο πολύπλοκος αυτός μηχανισμός διόρθωσης είναι μια επιτυχία σε ό,τι αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί ως στοιχείο επιτυχίας και όχι ως απειλή. Η δημοσιονομική αυτή διόρθωση του 1,8 δισεκατομμυρίων που εφαρμόστηκε στην Ισπανία το 2012 έχει να κάνει με δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις, με δύο συγκεκριμένους μάλλον λόγους διόρθωσης και έχει να κάνει και με θέματα ερμηνείας. Η ερμηνεία του άρθρου ε, του κανονισμού 438 του 2001 σε σχέση με την έκταση των προτέρων ελέγχων από τη διαχειριστική αρχή και δεύτερον η ερμηνεία των ευρωπαϊκών ε, οδηγιών σε σχέση με την ε, σύναψη συμβάσεων σε ό,τι αφορά τις δημόσιες συμβάσεις της χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά από πολλά χρόνια λοιπόν που εφαρμόζαν οι Ισπανικές αρχές κριτήρια και ερμηνείας που είναι γνωστές από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από την επιμονή της ίδιας ε, Εκτελεστικής Επιτροπής αλλάξαμε και τα κριτήρια και τις ερμηνείες και κάναμε ό,τι ήταν πιο δυνατό για να μπορέσουμε να εξαλείψουμε όλες τις ε, μορφές δαπανών που φυσικά ήταν απόλυτα νόμιμες στην Ισπανία αλλά δεν ε, συνάδουν με τις νέες ερμηνείες και τα κριτήρια της ε, Κομισιόν. Όλα αυτά ήταν δυνατό χάρη σε μια τεράστια προσπάθεια που κατεβλήθη από την Ισπανία τα τελευταία χρόνια και που ε, ουσιαστικά έπρεπε να αλλάξουν ένα μεγάλο μέρος του πλαισίου που έχει να κάνει με τις κοινωνικές δαπάνες. Δεύτερον, η μεγάλη ευελιξία που έδειξαν οι διαχειριστικές αρχές της Ισπανίας, οι οποίες ενώπιον ε, αλλαγών απότομων όπως αυτές που ε, που ζήτησε η Κομισιόν μπόρεσαν να αντιμετωπιστούν με τον πιο γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο και να προσαρμόσουν τη λειτουργία τους. Τρίτον, πρέπει να σταθώ στη διαφάνεια της διαδικασίας. Η έλεγχη του άρθρου 4 του κανονισμού 438 είναι κανονισμοί που έχουν να κάνουν αυτό που ονομάζουμε πολλές φορές εσωτερική κουζίνα των κρατών μελών και δεν υπάρχει υποχρέωση κοινοποίηση στην Κομισιόν, γιατί έχουν να κάνουν με την εθνική διαχείριση των λειτουργικών προγραμμάτων. Στην περίπτωση που μας ενδιαφέρει, η Κομισιόν πήρε πλήρη και λεπτομεριακή πληροφόρηση για όλες αυτές τις διαδικασίες που, όπως είπα προηγουμένως, έχουν εθελεντικό χαρακτήρα. Και γι' αυτό έχουμε τα ποσά αυτά τα οποία αναφέρθηκαν. Τέλος, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι με βάση την κρίση της ίδιας της Κομισιόν σε σχέση με τη διαδικασία αυτή, που έχει να κάνει με την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Η προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν πάντα η μέγιστη δυνατή. Υπήρξε διπλασιασμός των συστημάτων ελέγχου, ξεκινώντας και με το αρχικό σύστημα που εφήρμοσε η Κομισιόν και μετά με το τελικό το οποίο πρότεινε η Κομισιόν να εφαρμοστεί σε ό,τι αφορά την προστασία των κονδυλίων. Τώρα για την περίοδο 07-13. Δεν θα σας πω βέβαια ότι δεν είχαν προβλήματα. Είναι προφανές ότι τα δύο σημαντικά προβλήματα της περιοδου του 2000-2006 τα ξεπεράσαμε και τα συστήματα ελέγχου και τα νέα συστήματα για τις δημόσιες συμβάσεις ε, έχουν εφαρμοστεί με ικανοποιητικό τρόπο και αυτό το αναγνωρίζει και η Ισπανία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, έχουμε ένα σύστημα διαχείρισης και ελέγχου που έχει δυσκολίες προσαρμογής στις νέες προτεραιότητες και στα νέα προγράμματα. Από ένα μέσο επίπεδο χρηματοδότησης περίπου εκατομμυρίου σε ένα επίπεδο χρηματοδότησης που μόλις και μεταβία στάνει στις 100.000 ευρώ. Αυτό τι σημαίνει, ότι στην περίοδο 7-13 η Ισπανία χρειάστηκε να ελέγξει πάνω από είχε να ελέγξει καλύτερα πάνω από 300.000 ε, προσπάθειες, 300.000 ε, προγράμματα και πάνω από 10 εκατομμύρια ε, τιμολογίων. Ήταν λοιπόν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Ιδίω για τις υποδομές των μεταφορών και του περιβάλλοντος. Και εδώ είχαμε προβλήματα. Γιατί είχαμε τόσο πολύ περισσότερους ελέγχους να κάνουμε. Και οι έλεγχοι όχι μόνο δεν είχαν προσαρμοστεί στην αλλαγή τρόπο λειτουργία, αλλά συνέχισαν να χρησιμοποιούν μεθόδους που δεν ήταν τόσο αποτελεσματικέ για τέτοιου τύπου προγράμματα. Τα νέα συστήματα βασίζονται σε στάνταρ κόστος και προσπαθούν να ελέγξουν το αποτέλεσμα ή σε μεθόδους απλοποιημένου κόστου. Αυτά τα συστήματα άρχισαν να εφαρμόζονται μόνο στο τέλο περίοδου. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε περισσότερη προσπάθεια και την κάνουμε. Επίσης, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η αποκεντρωμένη ισπανική διοίκηση επίσης δεν ε, μας διευκόλυνε. Τώρα έχουμε πάνω από 150 ενδιάμεσους οργανισμούς που είναι επιφορτισμένοι με την διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης ε, ε, περιφερειακών πόρων και πάνω από 2.000 δικαιούχους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε μόνιμα μια προσπάθεια ελέγχου. Και όντω την κάνουμε. Και έχουμε δεσμευθεί ότι θα συνεχίσουμε να την κάνουμε. Τέλο. Δεν χρειάζεται να σα θυμίσω ότι η οικονομική κρίση στην οποία είμαστε βυθισμένοι και τα ασυμμετρικά αποτελέσματά της ε, στι χώρε τη Νότιας Ευρώπη σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε τεράστιες προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης που περιπλέκουν ε, τρομερά τόσο τη δυνατότητα εθνικής συγχρηματοδότησης, όσο και τη διατήρηση των υλικών και ανθρωπίνων πόρων που είναι αναγκαίοι για να υπάρχει σωστή διαχείριση, έλεγχος και επιθεώρηση της χρήσης των φόντων. Τώρα, για το μέλλον. Πρέπει να μάθουμε από το παρελθόν. Και η Ισπανία απέδειξε ότι μπορεί να προσαρμοστεί με ταχύτητα και ευελιξία στις νέες απαιτήσεις. Είναι προφανές ότι οι νέοι κανονισμοί, οι νέες προκλήσεις, δύσκολες σε πολλές περιπτώσεις. Θέματα όπως ε, η εξάντε ερεσιμότητα, η θεματική συγκέντρωση, οι νέες προτεραιότητες, η μείωση, για παράδειγμα, των εκπομπών ε, ε, οξυδίων άφρακα. Όλα αυτά δεν θα μας διευκολύνουν. Αντίθετα, μάλιστα. Στόχος μας, ωστόσο, είναι να ανταποκριθούμε όπως πάντα έχουμε επιχειρήσει. Να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις ταχαίως, με ευλίγιστο και διαφανή τρόπο. Για παράδειγμα, εργαζόμεθα σκληρά για να απλοποιήσουμε τα συστήματα ελέγχου, για να περάσουμε από αυτούς τους πάνω από 150 ενδιάμεσους οργανισμούς που προανέφερα, σε το πολύ 10 οργανισμούς δηλαδή συν 1 για κάθε αυτόνομη κοινότητα, δηλαδή 10 με 10 συν 17, 27. Νέες μεθόδους δηλαδή διαχείρισης που να προσαρμόζονται στα νέα χρηματοδοτικά μέσα, ιδιαίτερα όσον αφορά την ε, συγκεντρωτική διαχείριση, ιδιαίτερα για τα λειτουργικά προγράμματα. Να μην πω πολλά περισσότερα, για να μπορέσω να έχω χρόνο να απαντήσω και στις ερωτήσεις σας. Αλλά επαναλαμβάνω, ότι κάτω από κάποια στοιχεία που μπορεί να φαίνονται ε, αρνητικά ε, κρύβονται πολλές ε, περιπλοκότητες της κατάστασης αλλά εξακολουθούμε να εργαζόμεθα ούτως ώστε στο μέλλον να αλλάξει η κατάσταση και να καταλήξουμε σε μια πιο αποτελεσματική χρήση και μια διαφανή χρήση των ενωσιακών πόρων και ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Φερνάντες Κούρας, να ε, δώσω τώρα το λόγο στα μέλη για ερωτήσεις, να επενθυμίσω ότι επειδή πρέπει να αποφασίσουμε και για την απαλλαγή, ε, πρέπει να είμαστε ε, περιορισμένοι με το χρόνο. Λοιπόν, η Φιλία πρώτα, μετά Γκάια, μετά με συγχωρείτε, Τσαπατίνι, και, και ο Βόν, και ο, ο κύριος Ντέρεκ Βόν και η κυρία Γκρέσλε βεβαίω, Παρακαλώ. Ο κύριος Εφάτη, Η κυρία Εφάτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να χαιρετήσω την, τον κύριο Επίτροπο, τα μέλη του Ελεκτικού Συνεδρίου και προφανώς την ε, Υφυπουργό της Ισπανικής Κυβέρνησης που είναι παρούσα. Θέλω να την ευχαριστήσω και να την συγχαρώ για την παρέμβασή της που ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστική και μας έδωσε πολλά στοιχεία τα οποία μπορούν να μας οδηγήσουν σε καλύτερη κατανόηση της κατάστασης. Ενώπιον τώρα των διαφορών που υπήρξαν μεταξύ των Ισπανικών αρχών και των θέσεων του Ελεκτικού Συνεδρίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται η ανάγκη να υπάρξει μια συνεχής αλλαγή είτε σε διαδικασίες, είτε σε εφαρμογή των κανόνων και φυσικά και αλλαγή προτεραιότητων λόγω της οικονομικής κρίσης. Όλα αυτά μας υποχρεώσαν να, να τροποποιήσουμε την στάση μας στα θέματα αυτά στην Ισπανία. Θέλω να κάνω ε, μερικές ερωτήσεις σε σχέση με αυτά που είπατε κυρία Υπουργέ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αναφερθήκατε στην αλλαγή μεθοδολογίας που έπαιξε σημαντικό ρόλο. Θα ήθελα να μου δώσετε πιο συγκεκριμένα στοιχεία, αν μπορείτε, σε τι ακριβώς ε, συνίσταται αυτή η αλλαγή μεθοδολογίας που έχει πια οριστικό χαρακτήρα και επίσης αναφερθήκατε σε διαφορά, στη διαφορετική ερμηνεία του άρθρου 4 του κανονισμού 438 κάθετος 2001 για την εκ των προτέρων ε, εποπτεία και θα ήθελα να αναφερθείτε περισσότερο για το θέμα αυτό και επίσης θα ήθελα να αναφερθείτε αν θέλετε στις αλλαγές για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η συγχρηματοδότηση που αναφερθήκατε που και αυτές πιστεύω έχουν σημαντικό ρόλο στα αποτελέσματα που απεικονίζουν οι εκθέσει τη Κομισιόν και του Ελεκτικού Συνεδρίου. Σας προτείνω να συγκεντρώσουμε τις ερωτήσεις πρώτα για να πρώτο απαντήσετε. Ο κύριος Γκάιερ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υφυπουργέ, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την παρουσία σας. Αυτό είναι κάτι το οποίο το εκτιμούμε ιδιαίτερα. Το γεγονός ότι έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις με για την ε, εφαρμογή των διαφορετικών ταμείων στην Ισπανία. Ήμουνα το πες το καλοκαίρι στην ε, Μάλαγα, στην Ισπανία και νομίζω ότι έχω φτάσει σχεδόν στο σημείο που θα μπορούσα να μιλήσω εν μέρη την μητρική σας γλώσσα, αλλά έχω δει πολλά πράγματα για, τη λειτουργία των διαφορετικών πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μάλαγα. Είναι σαφές ότι υπήρξε κάποια βελτίωση και αυτό ως Ευρωβουλευτής μόνο χαρά μου δίνει. Δεν μπορώ να παραμεκφράσω την ικανοποίησή μου. Φυσικά, η χρηματοδότηση αυτή εξυπηρετεί και κάποιους πολιτικούς ε, στόχους όπως φάνηκε με τη δημιουργία πολιτιστικών κέντρων και του νέου ε, διαδρόμου περιπάτου στην Μάλαγα. Είχα την ευκαιρία να συζητήσω με τους εκπροσώπους των τοπικών αρχών, των αυτονόμων αρχών και συζητήσαμε για το τι μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των ε, αρχών, των θεσμικών αρχών, γιατί φυσικά τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία δαπανούν το 80% του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε κοινό συμφέρον να μειώσουμε το ποσοστό σφαλμάτων. Και φυσικά είμαστε υποχρεωμένοι να βλέπουμε σε ποια κράτη είναι καλύτερα, καλύτερη η εξέλιξη και σε ποια είναι λιγότερο καλή η εξέλιξη ποια είναι τα κράτη τα οποία πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια για να μπορέσουν να μειώσουν το ποσοστό σφαλμάτων. Και δυστυχώς η Ισπανία ε, είναι μία από τις χώρες όπου σε σχέση με τα διαφορετικά ταμεία υπάρχουν προβλήματα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη βελτίωση ίσως των πρακτικών της Κομισιόν, αλλά φυσικά από την άλλη πλευρά έχει να κάνει με την πολύπλοκη δομή που υπάρχει στη χώρα σας, γιατί οποιαδήποτε δαπάνη κονδυλίων πρέπει να γίνει μέσα από μια σειρά υπηρεσιών που είναι αρμόδιες στη χώρα σας, συναρμόδιες κατά κάποιο τρόπο λόγω των διαφορετικών επιπέδων και όταν πρέπει να περάσει 38 επίπεδα μια ε, εφαρμογή κονδυλίων, αυτό είναι φυσικό να οδηγεί και σε προβλήματα. Ελπίζουμε λοιπόν θα μπορέσει να δημιουργηθεί μια πιο απλή διαδικασία η οποία θα οδηγήσει σε λιγότερα σφάλματα, αλλά οι νέες δομές δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί από τη μια μέρα στην άλλη. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν η κεντρική κυβέρνηση στην Ισπανία πώς θεωρεί ότι θα πρέπει να διαμορφωθούν αυτές τις νέες δομές, τι σκέφτεται για την καλύτερη εκπαίδευση και κατάρτιση των δημοσίων υπαλλήλων στον τομέα αυτό και πόσο αισιόδοξοι μπορείτε να είσαστε ότι μπορεί έτσι να τροποποιηθεί η κατάσταση, αν το πω αλλιώ, πόσο γρήγορα νομίζετε ότι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε να υπάρξει σημαντική μείωση του ποσοστού σφαλμάτων στην Ισπανία. Και επομένως πόσο χρόνο, αν μπορείτε να το εκτιμήσετε, θα χρειαστεί για να ρονταριστούν κατά κάποιο τρόπο αυτές τι νέες δομές. Ευχαριστώ πολύ. Αράνκο. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Με βάση τις ε, οδηγίες σας που νομίζω ότι είναι πολύ καλές, ευχαριστώ την Υφυπουργό για την πληροφόρηση που μας έδωσε. Θα ήθελα να ζητήσω μια συμπληρωματική, ένα συμπληρωματικό στοιχείο γιατί δεν άκουσα να αναφερθήκατε σε ένα θέμα που νομίζω πως είναι σημαντικό. Δηλαδή, η εφαρμογή της γεωργικής πολιτικής, ιδιαίτερα μετά τη μεταρρύθμιση του 2015 για τις άμεσες πληρωμές. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει σωστή ε, καταγραφή των αγροτεμαχίων. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω εάν μπορέσετε να μας πείτε κάτι περισσότερο για το θέμα αυτό. Να μας πείτε τι προβλήματα έχει αυτό το σύστημα καταγραφής των αγροτεμαχίων και πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί αυτό το σύστημα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η συνάδελφος Γκρέσλε. Ναι, χαιρόμαστε πολύ που όντως ε, κάνατε ό,τι μπορούσατε για να μας ενημερώσετε. Να αναφερθώ στις ερωτήσεις ε, του εισηγητή. Συγκεκριμένα αυτό που υπόθηκε ότι όπως λέει και το συνέδριο 60% των σφαλμάτων θα έπρεπε να τα έχουν διαπιστώσει τα ίδια τα κράτη-μέλη. Ποιο είναι το πρόβλημα λοιπόν. Βεβαίως, καλά είναι όλα αυτά που μας λέτε, αλλά για την ε, ανάπτυξη και την απασχόληση αυτό δεν μας ε, προχωράει. Θα ήθελα να μας πείτε πώς εκτιμάτε εσείς ε, τα αποτελέσματα στην ανάπτυξη, και την απασχόληση των προγραμμάτων που εφαρμόζονται στην Ισπανία. Και θα ήθελα να μάθω να μας πείτε πώς μπορεί να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το κράτος μέλος της Ισπανία. Και συγκεκριμένα, τι θα κάνετε για να βοηθήσετε περαιτέρω την ε, διοίκηση στην Ισπανία. Βεβαίως, είναι περίπλοκο θέμα γιατί έχει να κάνει και με τη συνταγματική δομή της χώρας. Αλλά δεν θα έπρεπε και η πίεση που σας ασκούμε να σας βοηθήσουν να ε, εξυγχρονίσετε διοικητικές δομές που έχετε εδώ και δεκαετίες αν όχι αιώνες. Ευχαριστώ. Αγιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ και εγώ ευχαριστώ την Υφυπουργό για την παρουσία της που ανταποκρίθηκε δηλαδή στο αίτημα της Επιτροπής μας και συγκεκριμένα του εισηγητή και επαναλαμβάνω ότι υπήρξαν προβλήματα λόγω του ότι ακυρώθηκαν κάποιες πιστώσεις και μάλιστα σε κάποια τέτοια περίοδο. διότι υπήρξε και από τη δική μας τη μεριά του Κοινοβουλίου προσπάθεια να αναθεωρήσουμε τις μορφές χρηματοδότησης λόγω της κρίσης. Και το συνέδριο μας υπενθυμίζει ότι για κάποια προγράμματα του Κοινωνικού Ταμείου για την απασχόληση είχαν ζηθεί πριν από την κρίση ορισμένε συνθήκε. Για παράδειγμα, διατήρηση της ε, απασχόλησης για 3-4 χρόνια, αλλά κατόπιν ήρθε η κρίση. Και λόγω των απαιτήσεων ναι, για να υπάρξουν περικοπές και μεταρρυθμίσεις από πλευρά της Τρόικα, οι επιχειρήσεις δεν μπορούσαν να ε, συνεχίσουν με τον ίδιο αριθμό εργαζομένων. Άρα τις ίδιες αυτές τις συνθήκες χρειάστηκε να τις αναθεωρήσουμε. Το τονίζω και αυτό, γιατί και αυτό εξηγεί τι συνέβη και τι συμβαίνει ακόμη, τι δραματικά γεγονότα. Βεβαίως, αρχίσαμε να εφαρμόζουμε προγράμματα ανάπτυξης και απασχόληση, αλλά μετά ήρθε η κρίση. Και μας επέβαλε η Τρόικα συνθήκες ε, και ακριβώ αυτές τι συνθήκε εξετάζει αυτή τη στιγμή το Κοινοβούλιο εάν ήταν σωστές. Εφαρμόζονταν λοιπόν προγράμματα αλλά δεν μπόρεσαν τελικά να εφαρμοστούν σωστά και να διατηρήσουν ε, την απασχόληση. να διατηρήσουν την απασχόληση οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στα προγράμματα. Το διευκρινίζω αυτό γιατί τέθηκαν κάποια ερωτήματα. Γιατί τα θέματα αυτά κύριε Φιμπουργέ τα έχουμε συζητήσει και το ξέρουν όλοι οι συνάδελφοι. Άκουσα κάποια σχόλια και θέλω να σας ρωτήσω κύριε Υφυπουργέ. Όλοι αυτοί οι οργανισμοί ελέγχου που προσπαθείτε να μειώσετε Βεβαίω ξέρουμε ότι και σε άλλε χώρε υπάρχουν τέτοιοι οργανισμοί και γίνονται παρόμοιε προσπάθειε. Το είπε ο κ. Πίπερ για τη Γερμανία. Με τι τρόπο προσπαθείτε να βελτιώσετε την κατάσταση. Και δεύτερον, είπατε ότι μειώθηκαν οι πιστώσει. Μάλλον ε, ε, ανεστάλησαν πιστώσει για κάποιου τομεί, αλλά μπορέσατε κάποιε από αυτέ τι πιστώσει να τι αξιοποιήσετε αλλού. Αλλά συνολικά ποιο είναι το αποτέλεσμα για αυτές τι αναστολές ποιο πληρώνει τελικά οι Ισπανοί φορολογούμενοι και τι επίπτωση έχει στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Τι επίπτωση έχει αυτή η ακύρωση, η αναστολή προγραμμάτων. Ευχαριστώ. Ο Ντέρεκ Βόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την κυρία Υπουργό. Το 2012 εγώ ήμουν επικεφαλής μιας αντιπροσωπείας από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού στην Ισπανία και θυμάμαι ότι πολλοί πολιτικοί είπαν ότι ήρθαν κάποια σκοτεινά σκούρα κουστούμια που ήρθαν να μας πούν τι να κάνουμε. Βέβαια υπήρχαν και πολλές γυναίκες. Ε, δεν υπήρχαν πολλές γυναίκες σε αυτή την αντιπροσωπεία και εγώ φορούσα το ίδιο κοστούμι σε όλη την αντιπροσωπεία. Αλλά πήγαν παραγωγικά να επισκεφτούμε διάφορα σχέδια το τρένο υψηλής ταχύτητος, πήγαμε από τη Μαδρίτη στη Βαλένθια και επανήλθαμε. Είδαμε πολλά εγχειρήματα και σχέδια σε σχέση με, την, ε, τα συνδρομικά. Βέβαια συζητήσαμε και τις αναστολές και τις δημοσιονομικές διορθώσεις. Ένα σαφές και συνεχές επανερχόμενο θέμα ήταν αυτό με τον αριθμό των 150 ενδιαμεσών φορέων που εμπλέκονται στη χρηματοδότηση. Και χαίρομαι πάρα πολύ που λέτε ότι θα το μειώσετε από 150 σε 27. Αυτά είναι πολύ καλά νέα. Το ερώτημά μου λοιπόν περιστρέφεται γύρω από αυτό το θέμα. Για τα 27 αυτά νέα σώματα, νέους φορείς, μπορείτε να μας δώσετε κάποιες περισσότερες πληροφορίες πώς επιλέγονται, αν βασίζονται σε γεωγραφική κατανομή ή σε τομείς ε, δραστηριότητες, πώς λοιπόν θεωρείτε ότι μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση σε ό,τι αφορά την, ε, λειτουργία της, ε, την λειτουργία των χρηματοδοτήσεων. Ευχαριστώ. Τελευταίος, ο κύριος Γκαρίγα Πογέδο έχει το λόγο. Και ζητώ να λάβετε υπόψη και το χρόνο που περνάει. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Δύο ερωτήματα έθεσε ο κύριος Βον, ο οποίος ήταν επικεφαλής αντιπροσωπείας της Επιτροπής μας που μετέβη στην Ισπανία. Ε, ένα από τα θέματα που ετέθησαν κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης ήταν η συνεχιζόμενη <clears throat> αντίφαση μεταξύ του, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και της ισπανικής νομοθεσίας σε ό,τι αφορά τις δημόσιες συμβάσεις και την, τις τροποποίησεις που επήλθα. Θα μπορούσε τώρα η κυρία Υφυπουργός να μας εξηγήσει ποιες ήταν οι αλλαγές που έγιναν, τα μέτρα που ελήφθησαν από το 2012 για να υπάρξει περαιτέρω προσέγγιση μεταξύ των δύο νομοθεσιών. Δεύτερον, θα ήθελα, ατενίζοντας περισσότερο στο μέλλον, να έχω την ε, άποψη της ε, κυρίας Υφυπουργού για τον, ε, το πώς θα εφαρμοστούν οι νέες αυτές καθαρές δημοσιονομικές διορθώσεις σε διάφορα επίπεδα 5, 10 κτλ. Αν θεωρείτε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί και από τις εθνικές αρχές ελέγχου. Ευχαριστώ. Πάρα πολλά ερωτήματα, μια μεγάλη δέσμη ερωτήσεων και ελάχιστος χρόνος. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω ή δυνατόν σε 10 λεπτά να συζητήσετε γιατί να τα, να τα αντιμετωπίσετε γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε και το θέμα της ε, απαλλαγής 2012 εάν δεν μπορείτε και εγγράφως μπορείτε να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ λέει η κυρία Κουράνς. Θα προσπαθήσω να περιοριστώ στο χρόνο που μου δίνετε. παρά το γεγονός ότι πράγματι όπως είπατε είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί και είναι κεφαλαιόδους σημασία για τη χώρα μας. Πρώτα απ' όλα για την αλλαγή μεθοδολογίας. Θα πρέπει εδώ να σταθώ σε ένα θέμα το οποίο στην αρχή φαίνεται ότι είναι θέμα μονάχα ορολογίας. Ε, μίλησα για εθελοντικές ενέργειες είναι τα αποτελέσματα ενεργειών που έχουν γίνει από τις ίδιες τις διαχειριστικές αρχές. Κατά τη διάρκεια δηλαδή των προγραμμάτων που εφαρμόζονται, η Κομισιόν έχει διαπιστώσει ότι θα ήταν καλύτερη μια μορφή προληπτικού ελέγχου από αυτή που όπως έγινε και μετά από το 2006 και η Ισπανία απεδίθη σε μια εντυπωσιακή άσκηση διαθεσιμότητος, καλής πίστης, οργάνωσης, ευελιξίας για να υπάρξει καλύτερη προστασία των κοινωνικών, των κοινωτικών κονδυλίων, των ενωσιακών κονδυλίων. Ε, υπήρξαν μετά από το 2006 κάποιες διορθώσεις οι οποίες επιβεβαιώθηκαν. Δεν ήταν το 2012 που έγινε κάτι τέτοιο. Ήδη το 2011 είχαμε μονάχα 50 εκατομμύρια τα οποία αφορούσαν αυτές τις αλλαγές και αφορούσαν μονάχα τις διορθώσεις που είχαν στην πράξη εφαρμοστεί. Οι δύο μεθοδολογίες βέβαια έχουν και την δική τους καθεμία το τα δικά τους πλεονεκτήματα και τα αρνητικά τους. Θα ήταν χρήσιμο να έχουμε μια μεγαλύτερη προβλεψιμότητα και να μπορούμε να ξέρουμε ότι μιλάμε ακριβώς για τα ίδια πράγματα μέσα στο ίδιο χρονικό ορίζοντα. Το σίγουρο είναι ότι οι διορθώσεις οι οποίες επευλήθηκαν έχουν συσσωρευτεί και έχουν διογκωθεί τεχνικά ώστε όλα αυτά τα, όλες αυτές οι διορθώσεις οι οποίες αφορούσαν το διάστημα 2000-2006 εμφανίστηκαν σε μία μονάχα χρονική στιγμή. Το 1,8 δισεκατομμύρια που εμφανίστηκε το 2012 είναι το ποσό το οποίο έχει να κάνει με, το, με ένα σύνολο εκθέσεων που έτυχαν επιβεβαίωσης. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία μεταξύ του 2006 και του 2012 εμφανίστηκαν σταδιακά. Όλα αυτά λόγω της αλλαγής μεθοδολογίας για την ερμηνεία του άρθρου 4 και τους ελέγχους εξάντε που προβλέπει ο κανονισμός 438 του 2001 και θα πρέπει να πω ότι πέρσι το τελευταίο χρόνο μάλλον της περίοδου 2000-2006 η Κομισιόν έκανε κάποιες προτάσεις τροποποίησης σε σχέση με την ένταση των ελέγχων που έπρεπε να γίνεται από τους διαχειριστικούς φορείς. Η Γενική Διεύθυνση για τα κοινοτικά κονδύλια άρχισε να εργάζεται αμέσως, άλλαξε την, ε, τα κριτήρια που εφαρμοζόταν και φυσικά η ίδια αλλαγή έπρεπε να γίνει και σε όλες τις περιφερειακές διοικήσεις διαχείρισης Όλα αυτά λοιπόν έγιναν εκ των προτέρων προτού παρουσιαστούν οι ελτήσεις για καταβολή αποζημιώσεων και αυτό εφαρμόστηκε κατά 100%. Είναι γεγονός και πρέπει να το ομολογήσω ότι η Ισπανία δεν συμμεριζόταν απόλυτα την ερμηνεία της Κομισιόν σε σχέση με το άρθρο 4 και του κανονισμού 438. Δεν θεωρούσε ότι ήταν απαραίτητο να γίνουν όλα αυτά, αλλά συγχρόνως θα πρέπει να δεχτούμε ότι δεν θέλαμε να υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία σε σχέση με την αιρεσιμότητα των δικαιούχων που, και των κονδυλίων που δαπανήθηκαν από την Ισπανία. Τα πρώτα πέντε χρόνια της περίοδου 2000-2006 η Κομισιόν δεν είχε διατυπώσει καμία αντίρρηση για τον τρόπο με τον οποίο είχαμε λειτουργήσει. Και γι' αυτό το λόγο το πιο δύσκολο και οδυνηρό για μας και αυτό το οποίο θέλω να εξάρω είναι ότι κάναμε αυτές τις απαραίτητες ενέργειες σε ένα χρόνο ρεκόρ και με αναδρομικό χαρακτήρα εφαρμογής. Θα θέλαμε λοιπόν από αυτή την άποψη να τονίσουμε ότι για το μέλλον θα θέλαμε όλοι να κινούμε από κοινού και να μπορέσουμε να γνωρίζουμε ποιες είναι αυτές οι αλλαγές γιατί ανεξάρτητα από τη μορφή που έχει η διοικητική οργάνωση μιας χώρας είναι πεπερασμένη η ικανότητα αντίδραση σε απότομες αλλαγέ. Η Ισπανία είναι η τέταρτη οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό σημαίνει ότι ε, χρειάζεται να καταβάλουμε μια εξαιρετική προσπάθεια για να κάνουμε αυτές τις αλλαγές και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να κάνουμε τις απαραίτητες προσπάθειες εάν θεωρείτε ότι δεν έχουν αντιμετωπιστεί πλήρως όλα αυτά τα θέματα. Ελπίζουμε ότι θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε τόσο, σημαντικά, ε, τόσο σημαντικές αλλαγές σε αναδρομικό επίπεδο. Ε, θα ήθελα επίσης να σας τονίσω ότι η Ισπανία είναι μια χώρα η οποία από τη στιγμή της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σταθεί ένας από τους μεγαλύτερους δικαιούχο, δικαιούχους ε, διαρθωτικών πόρων που έπαιξαν κατά κάποιο τρόπο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην οικονομία της Ισπανίας, οδήγησαν σε μια σημαντική αύξηση του μέσου κατακεφαλή εισοδήματο στην Ισπανία και είχαν μια ιδιαίτερη προσθέμενη αξία ότι έδωξαν τον ρόλο υποδείγματος και οδηγού για την σωστή για τις σωστές ε, επενδύσεις, τις ε, εποφελείς επενδύσεις που θα μας οδηγούσαν σε μια μεγαλύτερη σύγκληση και προσέγγιση στους Ευρωπαίους μας εταίρους. Θεωρώ ωστόσο ότι η Ισπανία ίδια ως κράτος έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια επενδύσεων. 15% είναι οι ενωσιακοί πόροι, 85% είναι ήδη οι πόροι εθνικοί. Και ο συνδυασμός αυτών των δύο βεβαίως είναι πολύτιμος. Η Ισπανία ήθελε πάντα να βοηθήσει την έρευνα και την ανάπτυξη. Και πάντα λαμβάναμε υπόψη ε, την διάσταση αυτή που μπορεί να σημαίνει ότι δεν λαμβάνει υπόψη όλες τις άλλες διαστάσεις. Αλλά βεβαίως οι διαφθορτικοί πόροι μας ε, βοήθησαν πολύ. Αλλά διάφορες ισπανικές κυβερνήσεις έκαναν μία μόνιμη προσπάθεια επενδύσεων που μας επέτρεψαν να έχουμε αυτήν την ευελιξία. Δηλαδή, ανα πάσα στιγμή, χάρη ε, στο ρόλο ε, ενάυσματος που μας έδινε η Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούσαμε εμείς με περισσότερη ευελιξία να παράσχουμε τη συμπληρωματική χρηματοδότηση. Έχουν γίνει πολλές ερωτήσεις που μπορώ να τις αντιμετωπίσω από κοινού γιατί βλέπω ότι υπάρχει κάποια ανησυχία για το πώς θα τα πάει και τι θα κάνει η χώρα μας για να βελτιωθεί η διαχείριση των πόρων. Θέλουμε να απλοποιήσουμε φυσικά τις διοικητικές μας ε, δομές. Ξέρετε ότι η χώρα μας έχει πολύ μεγάλο βαθμό αποκέντρωσης και σε μεγάλο βαθμό οι αυτόνομες κοινότητες ε, αναλαμβάνουν την ε, διαχείριση των πόρων και πολλές φορές και τοπικοί φορείς. Θέλω να τονίσω ότι η Ισπανική κυβέρνηση δεσμεύεται να απλοποιήσει και να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό. Διότι, βεβαίως, έχουμε μια συγκεκριμένη διοικητική και πολιτική ταυτότητα που απορρέει από το Σύνταγμά μας το 1978. Αλλά υπάρχει πολλή συνεργασία που θα μπορούσε να επιτευχθεί μεταξύ των ε, διοικήσεων για να βελτιωθεί η κατάσταση. Είμαι αισιόδοξη. Πιστεύω ότι, πιστεύω ότι αυτή η διαδικασία αναδιοργάνωσης γίνεται με βάση ένα πολύ φιλόδοξο πολιτικό στόχο που αφορά όλες μας τις εθνικές δομές. η κυβέρνηση έχει το εξή σύνθημα. Θέλει δηλαδή οι δομές μας να είναι απλές και να βασίζονται λοιπόν στην αρχή μία διοίκηση, μία αρμοδιότητα. Πολλές πολιτικές και κανονιστικές πρωτοβουλίες αναλαμβάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Για παράδειγμα, έχουμε την έκθεση Κόρα, που είναι μια έκθεση που προσπαθεί να αποφευθεί η διοικητική επικάλυψη σε διάφορους τομείς που προκαλεί ε, διαδικασίες ε, σπατάλησης ε, πόρων, χρόνου κτλ. Δηλαδή, πιστεύω ότι θα υπάρξει ικανοποιητική πρόοδος. Θέλουμε λοιπόν να υπάρξει μια κουλτούρα συντονισμού. Οπωσδήποτε θα την αξιοποιήσουμε για τη χρήση των ενωσιακών πόρων, συμπεριλαμβάνοντας τις προσπάθειες λοιπόν να ξεπεράσουμε αυτές τις, ε, αυτούς τους 150 φορείς ε, που θέλουμε να τους ε, αντικαταστήσουμε με το πολύ 27. 10 σε εθνικό επίπεδο όπως ακριβώς με ρωτήσατε, οι οποίοι θα φορούν συγκεκριμένους τομείς και 17 άλλους φορείς με βάση εδαφική κατανομή. Δηλαδή ένα τέτοιο φορέα ανά αυτόνομη κοινότητα. Πρόεδρος, σας παρακαλώ μήπως ε, να απαντήσετε ε, γραπτά στις υπόλοιπες ερωτήσεις γιατί δεν θα έχουμε χρόνο για την έκθεση απαλλαγής της Επιτροπής. Γιατί είχα, είχα προβλέψει για την εισαγωγική παρουσίαση τρία λεπτά, κράτησε 20 εισαγωγική παρουσίαση. Βεβαίω τέθηκαν πολλά ερωτήματα, μήπω θα μπορούσατε να απαντήσετε γραπτό παρακαλώ στα υπόλοιπα ερωτήματα. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε. Σας ευχαριστώ που ήρθατε να μας δείτε, κυρία Υπηφυπουργέ. και παρακαλώ να στείλετε γραπτή απάντηση στις επόμενες ερωτήσεις, στις υπόλοιπες ερωτήσεις. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν θα λάβει το λόγο για το θέμα αυτό η Κομισιόν. Να μας απαντήσει γραπτός και εκείνη. Και να περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα της μέρης διάταξης. Έκθεση απαλλαγής. Ο εισηγητής. Ευχαριστώ. Λοιπόν, και εγώ θα πω τα μισά από όσα προέβλεπα να πω. Ξεκινάω λοιπόν. Με κάτι που θα, ήθελα, θα θέλαμε τις τελευταίες εβδομάδες ε, να, μας, να έχει κάνει η Κομισιόν. Αλλά θα ξεκινήσω με έπαινο. Ακούσαμε για τα προβλήματα σε διάφορες ε, χώρες μέλη, δεν θα τα παραλάβω. Νομίζω ότι η Κομισιόν καταδεικνύει προβλήματα σε, διάφορες, ε, σε διάφορους τομείς, αναφέρεται στην έκθεση Γκάιερ και επαναλαμβάνει διάφορες προτάσεις. Θεωρούμε ότι είναι θετικό ότι οι μηχανισμοί επιβολής κυρώσεων στον γεωργικό τομέα και στον τομέα συνοχής θα εξομοιωθούν. Αυτό θα είναι δυνατό και για την περιφερειακή πολιτική με τις καθαρές οικονομικές διορθώσεις. Έχουμε δυνατότητα λοιπόν αναστολής και διακοπής ε, πληρωμών. Θα βελτιώσει την κατάσταση. Πολύ καλό επίσης ότι η έκθεση για την ε, προστασία των οικονομικών συμφερόντων τη Ένωση κάνει διακρίσει αναχώρε και αυτό είναι θετικό. Και επίση το πρόγραμμα δράση για την ανώδεξη τη υπαίθρου και αυτό το θεωρούμε θετικό και την αύξηση των τιμών κατοφλίων. Αυτό οπωσδήποτε θα οδηγήσει σε λιγότερα λάθη. Και τέλο, αλλά όχι και ασήμαντα. Βλέπουμε να υπάρχει και ή ακούμε να υπάρχει και ένα άτυπο χρονοδιάγραμμα πώ θα προσπαθήσει να υπάρξουν καθαρές οικονομικές διορθώσεις με ευθύνη της Κομισιόν. Θα έχουμε δηλαδή τους επόμενους μήνες μια πιο συγκεκριμένη εικόνα της κατάστασης. Όλα αυτά είναι πολύ θετικά. Αλλά, αλλά, ένα σημαντικό αλλά θα αναφέρω τώρα. Για μια διαδικασία απαλλαγής δεν υπαρκεί να βασιστούμε σε ελπίδες. Κάναμε επικρίσεις στο παρελθόν. Τώρα σε κάποιους τομείς ε, υπάρχουν κάποιες ε, προσπάθειες και να βασιστούμε λοιπόν σε αυτό για να δώσουμε 100% απαλλαγή δεν επαρκεί. Σε ορισμένους τομείς οι μηχανισμοί δεν είναι επαρκείς. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει συστηματική δειγματολοπτική προσέγγιση της Κομισιόν. Ακούσαμε ότι οι εκθέσεις ελέγχου από τις ε, χώρες μέλη δεν είναι επαρκής για να οικοδομηθεί επ' αυτόν ένα σύστημα ελέγχου. Γι' αυτό πρέπει να αναλάβει αυτοδέσμευση Κομισιόν που να μπορούμε να την παρακολουθήσουμε ότι αυτή η ίδια θα κάνει ελέγχους στους τελικούς δικαιούχους και στους οργανισμούς, τους εθνικούς που, κάνουν, που εγκρίνουν τις πληρωμές. Στους οργανισμούς που εγκρίνουν τις πληρωμές. Γιατί εδώ έγιναν τα λάθη στο παρελθόν. Εδώ έγιναν τα περισσότερα λάθη. Δεν όχι, αυτό δεν σημαίνει ότι χρειαζόμαστε περισσότερους ελέγχους, περισσότερη αυτοκρατία. Χρειαζόμαστε πιο στοχευμένους ελέγχους σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Θέλουμε λοιπόν να αναλάβει πρωτοβουλίες για αυτό η Κομισιόν. Τι άλλο περιμένουμε. Να περιοριστεί η αντικατάσταση προγραμμάτων. Νομίζουμε ότι οι πολύτιμοι πόροι σε πολύ μεγάλο βαθμό μπλοκάρονται. Μετά προκύπτουν διοικητικές διαδικασίες που δεν βλέπουμε τι στόχο έχουν. Και αυτό οδηγεί σε απώλειες στον προϋπολογισμό. Θα πρέπει να υπάρχει όριο για αυτήν την αντικατάσταση προγραμμάτων. Στη Γεωργία. Έχουν γίνει ήδη καθαρές ε, οικονομικές διορθώσεις, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και κυρώσεις. Όταν, χρόνο μετά το, δηλαδή όταν επανειλημμένα, χρόνο με χρόνο, ε, γίνονται διορθώσεις, τότε θα πρέπει να υπάρχει και σημαντική κύρωση, πρόστιμο, επιπλέον κάτι. Και αναφέρομαι ιδιαίτερα στο σύστημα για την καταγραφή των ε, αγροτεμαχίων. Δηλαδή, εάν κάθε φορά που παρκάρω παράνομα ε, πληρώνω πρόστιμο 5 ευρώ, θα συνεχίσω να το κάνω κάθε χρόνο, κάθε μέρα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να είναι κλιμακωτά αυτά τα πρόστιμα και αν συνεχίσει παρόλα αυτά η κατάσταση τότε θα πρέπει να το πάρει και ο Γερανός το αυτοκίνητο κάποια στιγμή. Παράλληλη λοιπόν πρέπει να είναι η κατάσταση. Αν δεν βελτιώνεται η κατάσταση, θα πρέπει η Κομισιόν να αναλαμβάνει περισσότερη άμεση ευθύνη. Αυτό είναι βασικό για μας. Και κάτι άλλο προς το ελεκτικό συνέδριο. Θα πρέπει να αντιδράσει επιτέλους και το ελεκτικό συνέδριο. Παρά όλα τα θετικά που μας έχει στείλει, όσο δεν υπάρχουν εκθέσεις για τις χώρες που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα προγράμματα, δεν θα μπορέσουμε να πάμε σε βάθος τον ελεγχό μας. Και αυτό είναι πολύ βασική απέτηση που σχετίζουν με την διαδικασία απαλλαγής. Κυρίες και κύριοι, είναι σαφές ότι κύριος στόχος της κριτικής μας είναι η αμελής χρήση των ενωσιακών πόρων σε ορισμένα κράτη-μέλη. Βλέπουμε ότι η αρχή της επιμερισμένης διοίκησης δεν πρέπει να τεθεί να αμφιβόλο γενικά. Κάποια κράτη-μέλη πρέπει να αμφισβητηθούν για το πώς ενεργούν. Γιατί κάποια κράτη-μέλη λένε καλά, ενωσιακή πόρη, εντάξει, μπορούμε να είμαστε χαλαροί. Αυτό στο μέλλον δεν πρέπει να συνεχιστεί. Δεν πρέπει. Και γι' αυτό εκφράζουμε επιφυλάξει για την γεωργία και την περιφερειακή πολιτική. Σε αυτού του τομεί έχουμε επιμερασμένη διοίκηση, επιμερισμένη διαχείριση. Και τονίζω ότι αυτές οι επιφυλάξεις πρέπει να απευθυνθούν με πολύ πιο βαρύ τρόπο προς τα κράτη-μέλη. Βεβαίως, η Κομισιόν είναι θεματοφύλαξη των συνθήκων. Αλλά εάν ε, δείξουμε κίτρινη κάρτα στην Κομισιόν, τότε πρέπει να δείξουμε μια βαθύ πορτοκαλιά κάρτα στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει οπωσδήποτε να συζητηθούν τα θέματα αυτά. Βεβαίω ξέρω ότι ε, υπάρχουν και ισχυρέ επικρίσει κατά των επιφυλάξεων. Αλλά τι θέλετε να κάνουμε. Με βάση τη συνθήκη Μπορούμε να πούμε μόνο ναι ή όχι στη διαδικασία απαλλαγή. Είτε δηλαδή θα πρέπει να ρίξουμε ατομική βόμβα ή να του χαϊδέψουμε. Αυτό έχει γίνει τόσα χρόνια όμω. Εντάξει, του αφήνουμε, τους αφήνουμε να περάσουν, του χαϊδεύουμε, ε, κάνουμε κάποιε επιφυλάξει και κανεί δεν ασχολείται με αυτέ. Πρέπει λοιπόν να αυτοδεσμευτεί και το Κοινοβούλιο να δει τι θέλει να επιτύχει με αυτές τις επιφυλάξεις. Να μην ξεχνούνται δηλαδή αυτές οι επιφυλάξεις. Και πριν επικρίνει αυτή την ιδέα η Κομισιόν, παρακαλώ και το συνέδριο να έχει πιο διαφοροποιημένη ε, αντιμετώπιση. Έχει διαφοροποιημένη γνώμη ανάλογα με τις ε, δαπάνες, τις, ε, τα έσοδα κτλ. Γιατί και η Κομισιόν να μην κάνει πιο διαφοροποιημένη ε, δήλωση αξιοπιστίας και αποδοχής. Να πούμε λοιπόν ότι αναμένουμε ότι έχουν αξιοποιηθεί σωστά επιστώσει για τα προγράμματα εκτός από εκείνα που η Κομισιόν έχει εγκρίνει με επιφυλάξει και παρατηρήσεις. Γιατί λοιπόν αυτές τις επιφυλάξεις να μην τις αξιοποιήσουμε πολιτικά, να είναι πιο συγκεκριμένη η προσέγγιση μας. Θα ήταν πολύ λογικό αυτό να το κάνουμε και το οποίο σημαίνει ότι αναλαμβάνουμε τι ευθύνε μα. Τώρα δεν θέλω να δημιουργήσω λάθος ε, εντυπώσεις. Ξέρω ότι υπάρχουν ε, φήμες ότι ε, δεν θα χορηγήσουμε απαλλαγή ή ότι θα αναλάβουμε την απόφασή μας. Όχι, δεν το λέει αυτό η έκθεσή μου. Καλό είναι να χορηγηθεί απαλλαγή. Αλλά χορηγούμε απαλλαγή με επιφυλάξεις που ελπίζουμε να μας επιτρέψουν στο μέλλον να ασχοληθούμε πολύ εντονότερα με τα θέματα αυτά. Αυτό θα πρέπει να γίνει αποδεκτό ότι πρέπει να το επιχειρήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ελπίζω να το αποδεχτούν και οι συνάδελφοί μου από τι άλλε πολιτικέ ομάδε και η Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σίγητα. Δίνω το λόγο στον Επιτροπό μας. Δεν χρειάζεται να τον παρουσιάσω. Βέβαια έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Ισηγητά για την παρουσίασή σας, κυρίες και κύριοι. Θέλω πρώτα να τονίσω ρητά ότι η Κομισιόν συμμερίζεται τις ίδιους στόχους με τον εισηγητή. Η Κομισιόν θεωρεί πράγματι ότι παρά τις προσπάθειες που έγιναν για να προστατευθεί αποτελεσματικά ο ενωσιακός προϋπολογισμός, ο ρυθμός λαθών πρέπει να μειωθεί. Τα τελευταία χρόνια η Κομισιόν εφάρμοσε έναν εντυπωσιακό αριθμό μέτρων, αλλά ο ρυθμός λαθών συνεχίζει αμύωτος. Άρα χρειάζεται περαιτέρω βελτιώσεις. Γιατί λοιπόν υπάρχει αυτή η κατάσταση το 12. Ας μην αναφερθώ εκ νέου στην αλλαγή της μεθοδολογίας του ελεγκτικού συνεδρίου. Θα ήθελα απλώ να τονίσω ότι το μεγαλύτερο τμήμα των λαθών ε, οφείλεται στα κράτη-μέλη λόγω της ε, κοινής διαχείρισης. Η επικουρικότητα δεν σημαίνει μόνο να λαμβάνονται αποφάσεις στο καταλληλότερο επίπεδο, αλλά σημαίνει επίσης να αναλαμβάνουμε πλήρως τις ευθύνες μας, τις ευθύνες που απορρέουν από τις αποφάσεις αυτές. Το λέει καθαρά το 317 της συνθήκης και ο, χρηματο... και ο δημοσιονομικός κανονισμός. Γι' αυτό η Κομισιόν θεωρεί ότι το να δοθεί κίτρινη κάρτα σε αυτήν με τη μορφή πολιτικών επιφυλάξεων όπως κάνει η εισηγητή είναι σαν να έδινε κίτρινη κάρτα στον ίδιο το διαιτητή χωρίς να τη δίνει στους παίκτες που παραβιάζουν τους κανόνες και γι' αυτόν τον λόγο εξήγησα ήδη προς τον εισηγητή ότι οι πολιτικές του επιφυλάξεις για το 17% του προϋπολογισμού ιδιαίτερα για την περιφερειακή πολιτική και τη γεωργία δεν επιτυχάνουν το στόχο που έθεσε αντίθετα αμφισβητούν την ε, νομιμότητα της Κομισιόν έναντι όλων των δημοσιονομικών και χρηματοπιστωτικών παραγόντων ενώ χρειάζεται άλλος τρόπος για να μειωθούν αποτελεσματικά τα λάθη. Ας έρθω τώρα στο σχέδιο απαλλαγής και τον τρόπο με τον οποίο θέλει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που ταυτίστηκαν οι Κομισιόν. Για τη νέα στρατηγική δημοσιονομικού ελέγχου έχω ήδη πει ότι θα υποβληθεί λεπτομεριακά για την επόμενη διαδικασία απαλλαγής, όπως λέει και το σχέδιο ψηφίσματος. Από το 9 τα διαρθρωτικά ταμεία και οι ανάλογες γενικές διευθύνσεις έχουν προσπαθήσει να ταυτίσουν ε, τις διαδικασίες εποπτείας και ελέγχου των εθνικών αρχών και κάλυψαν 47 περιφερειακά ταμεία και 85 κοινωνικά προγράμματα από τα κοινωνικό ταμείο και οι γενικές αυτές διευθύνσεις θα συνεχίσουν να αυξάνουν τις προσπάθειές τους με βάση την εμπειρία που έχουν αλλά και με την ταύτιση σημαντικών κριτηρίων κινδύνου ή αδυναμιών που θα έχουν ταυτιστεί από διάφορα, σε διάφορα κράτη-μέλη και θα γίνουμε αυστηρότεροι για την λήψη διορθωτικών μέτρων. Η Κομισιόν επίσης θα ακολουθήσει τη σύσταση να τους ελέγχους που κάνει, τους δηματοληπτικούς ελέγχους, με βάση την καινούργια μεθοδολογία. Τώρα όλα αυτά θα εφαρμοστούν και για την πολιτική συνοχή συστηματικά δηλαδή αδιάκριτα και με διαφανή κριτήρια όπως ορίζουν οι κατεξουσιοδότηση πράξεις. Οι διορθώσεις θα είναι ρεπτομεριακές και θα εμφαίνονται στην επόμενη ετήσια έκθεση. Η Κομισιόν θα εξετάσει πώς να βελτιώσει και την παρουσίαση που κάνει στην ετήσια έκθεση πεπραγμένων της για να συμπεριλαμβάνει σε αυτήν και πληροφορίες ως προς τη χρήση των πληροφοριών για την ανάλυση κινδύνου και τις δημοσιονομικούς ελέγχους που έχουν κάνει τα κράτη-μέλη που, από την οποία πηγάζει και η δική μας τελική μελέτη. Επίσης συμφωνούμε ότι οι διαδικασίες ε, συμμόρφωσης δεν πρέπει να ξεπερνούν τα δύο χρόνια θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Όσο για το πρόβλημα που ταυτίστηκε στη Γαλλία και την Πορτογαλία, που το αναφέρει και αυτό η έκθεση, το σχέδιο έκθεσης για τη Γεωργία, το σχέδιο δράσης για την Πορτογαλία έχει συμπληρωθεί και θα γίνει αξιολόγησή του όταν θα έχουμε τα στοιχεία των δημοσιονομικών ελέγχων. Για τη Γαλλία ένα σχέδιο δράσης έχει εγκριθεί από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας, αλλά απαιτεί ακόμη πολλή δουλειά από τις γαλλικές αρχές τα επόμενα χρόνια για να ενημερωθούν όλα τα στοιχεία που διαθέτουμε. Η, τα milestones θα τα εξετάσει η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας με το στόχο να γίνει ενημέρωση και εξυγχρονισμός των δημοσιονομικών ελέγχων. Επίσης πιστεύουμε ότι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους οι εθνικές αρχές διαχείρισης μέσω των σχετικών δηλώσεων που πρέπει να υποβάλουν κάθε φορά. Επίσης, είμαστε αποφασισμένοι να διευκολύνουμε και να προωθήσουμε τη χρήση εθνικών εθελοντικών δηλώσεων βάσει του προτύπου και των συστάσεων που θέσπισε η διαθεσμική ομάδα εργασίας. Τέλος, ένα καινούργιο πλαίσιο αποτελεσματικότητας έχουμε καθορίσει για να είναι όλα αυτά να καταλήγουν σε περισσότερη υπεραξία για τους πολίτες με συγκεκριμένους στόχους και δείκτες που θα εφαρμόζονται για όλες τις νομοθετικές πράξεις των συνομοθετών. Για τα έσοδα και τους ιδίους πόρους, τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους. Υπάρχει επίσης ένα σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαπάτης για τα τελωνία και τους δασμούς. Έχουμε επίσης προτάσεις για την καταπολέμηση και εκεί της απάτης μέσω ποινικών μέτρων. Από τον Ιούλιο του 12 το Συμβούλιο ενέκρινε το νέο μηχανισμό γρήγορης ανταπόκρισης για να μπορέσουμε έτσι να αντιμετωπίσουμε ξαφνικά προβλήματα που μπορεί να διαπιστωθούν στα κράτη-μέλη. Όσο για την ανατροπή των επιφυλάξεων για τα στοιχεία GNI και για τα στοιχεία της ΕΖΕΣ, θα σας τηρούμε ενήμερους. Τον Ιούνιο του 2013 η Κομισιόν επίσης ενέκρινε μια ανακοίνωση προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Αναβάθμιση του αντιμετώπιση του λεφρεμπορίου σιγαρέτων που αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει να εφαρμόζεται. Συμμερίζομαι τις ανησυχίες του εισηγητή ως προς την αναγκαιότητα να τα προσέχουμε όλα αυτά από κοντά για τα ράλι ιδιαίτερα. Γιατί ένας τέτοιος καλύτερος έλεγχος θα ταυτίσει ευκολότερα τα προβλήματα και εμείς είμαστε αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουμε αυτό το εργαλείο ελέγχου πιο συχνά. Όλα αυτά τα μέτρα που σας παρουσίασα κυρίες και κύριοι θα συμπεριληφθούν σε μια λεπτομερή επιστολή που θα σας έρθει τις επόμενες ημέρες στην Επιτροπή σας και αποδεικνύουν ότι είμαστε αποφασισμένοι στην Κομισιόν να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να εξηγήσουμε γιατί οι πολιτικές αυτές επιφυλάξεις που αναφέρει η συγητής δεν είναι σωστέ να αναφέρονται σε αυτή την έκθεση απαλλαγής. Η επιστολή αυτή ελπίζουμε ότι θα συμβάλλει σε πιο επικοδομητικά αποτελέσματα για τη διαδικασία απαλλαγής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πρώτα για τη δήλωσή σας. Και ξεκινάει η συζήτηση. Θα ήθελα καταρχήν να ξέρω ποιοι συνάδελφοι θα θέλαν να λάβουν το λόγο ώστε να καθορίσω καλύτερα το, την κατανομή του χρόνου. 20 λεπτά έχουμε μόνο. Δύο λεπτά στον κάθε ομιλητή τότε. Τέσσερα. Τέσσερις λοιπόν. Τρία λεπτά, τρία λεπτά, ναι. ναι. Ωραία. Ο Derek Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον Επίτροπο και τον εισηγητή για τη συμβολή τους στο θέμα αυτό. Είδαμε ότι υπήρξε αυτή η αύξηση φαλμάτων στα 4,8% και φυσικά είναι υπερβολικά ψηλό αυτό το ποσοστό. Ο κύριος Επίτροπος εξήγησε γιατί υπήρξε αυτή η αύξηση στο ποσοστό σφαλμάτων με τον ε, ε, κύριο λόγο να είναι η αλλαγή μεθοδολογία, αλλά οι, δια, οι διορθώσεις στα καταποκοπή ποσά ίσως δεν έχουν ληφθεί πλήρως υπόψη σε αυτήν την περίπτωση. Υπάρχουν επίσης πολλά μικρά προγράμματα τα οποία, στα οποία γίνονται καταβολές πληρωμών μόνο στο τέλος της διάρκειάς τους. Αλλά υπάρχει και το θέμα της ε, λειτουργίας των κρατών μελών για τα θέματα αυτά και χαίρομαι πάρα πολύ που ο εισηγητής το έχει αναγνωρίσει αυτό το θέμα. Υποστηρίζω πολλά από αυτά που λέει ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη επαρκούς ε, δράσεις για τα θέματα αυτά στα κράτη-μέλη και να θέσουμε περισσότερο την έμφαση στα προβληματικά κράτη-μέλη. Κάτι ακόμα όμως το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι η ιδέα αυτή των πολιτικών επιφυλάξεων που ανέφερε ο εισηγητής και αναφέρθηκαν και από τον Επίτροπο επίσης. Η ομάδα των σοσιαλιστών έχει πρόβλημα με κάτι τέτοιο. Είναι η πρώτη φορά που διατυπώνεται μια τέτοια ιδέα για μας Αυτό σημαίνει να αναβάλουμε την απαλλαγή μέχρι αργότερα το χρόνο και αυτό δεν προωθεί το διάλογο για τα κράτη-μέλη τα οποία δεν ε, τα οποία πρέπει να έχουν περισσότερη προσοχή. Είναι σαν να επιβάλλουμε κυρώσει στα αυτοκίνητα που είναι νόμιμα παρκαρισμένα, όπως θα έλεγε και ο εισηγητή. Επίση θα έχει επιπτώσει και για τα προγράμματα του 2014 και δεν μα δίνει επαρκή χρόνο να κατανοήσουμε αν όλες αυτές οι αλλαγέ έχουν οδηγήσει σε βελτίωση. Όσο δεν έχουν λοιπόν περατωθεί, όσο δεν έχει ε, περατωθεί η εφαρμογή αυτών των ε, σχεδίων που υπόκειται σε κατεξουσιοδότηση πράξη και δεν έχουν δοθεί οι απαραίτητε πληρωμέ, δεν έχουμε στην πραγματικότητα το χρόνο να δούμε κατά πόσο έχουν γίνει οι βελτιώσει και έχει επιτευχθεί η πρόοδο αυτή που θέλαμε να έχουμε. Και θεωρούμε ότι ίσω δεν έχει νόημα να θεωρήσουμε υπεύθυνο το νέο επίτροπο για την διαδικασία απαλλαγή του 2012. Θα πρέπει να επέχουν την ευθύνη για τα νέα προγράμματα, όχι για τα παλιότερα προγράμματα. Αντί λοιπόν να έχουμε αυτές τις πολιτικές επιφυλάξεις που αναφέρθηκαν, θα πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένες αιτήσει προς τα κρατημέλη, προς το ελεκτικό συνέδριο, αλλά και προς την Κομισιόν <clears throat> να εστιάσουν σε ιδιαίτερους τομείς όπου χρειάζεται περισσότερη πρόοδος στο μέλλον. Και μπορούμε να συζητήσουμε για ποιους τομείς θα πρέπει να αναφερθούμε να εστιάσουμε στα πιο ασθενή κράτη-μέλη και κατά πόσο θα πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο δράσης για τα πιο προβληματικά κράτη-μέλη, να έχουμε νέα εργαλεία συνοχής, ε, ε, να έχουμε ένα καλύτερο μηχανισμό συμψηφισμού των οφελών, οφειλών στη γεωργία, να έχουμε καλύτερη παροχή αναφορών, μια στρατηγική που να βασίζεται στην εκτίμηση κινδύνου για τους λογιστικούς ελέγχους. Να το τελειώσω αυτό κύριε Πρόεδρε. Αυτό που λέμε λοιπόν είναι ότι σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να δώσουμε την ε, απαλλαγή, αλλά να κάνουμε κάποιες επίσημες αιτήσει για περαιτέρω πρόοδο στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος Ντέρεκ είναι Σαγιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα και εγώ θέλω να υποστηρίξω αυτά που έλεγε ο Ντέρεκ Βόν και θέλω να ζητήσω από τον πρόεδρο της Επιτροπής μας και τα άλλα μέλη της Επιτροπής μας να ζητήσει από την νομική μας υπηρεσία μια γνωμοδότηση για τις επιφυλάξεις αυτές που αναφέρθηκαν. Γιατί η Κομισιόν ουσιαστικά βρίσκει όλο και περισσότερες, η Επιτροπή μας μάλλον, μπορεί να φανταστεί κάποια φόρμουλα για να δώσει, να μην δώσει την απαλλαγή και βρίσκουμε τρόπους να πούμε ναι μεν αλλά ή όχι μεν αλλά. Λοιπόν, οι φήμες κυκλοφορούν εδώ πέρα ε, για το τι θα κάνουμε, τι δεν θα κάνουμε, όλα αυτά δεν έχουν καμία ουσία σε νομικό επίπεδο. Δεύτερον, θα ήθελα να τονίσω τη ματέωση που νιώθω με τον κύριο Πίπερ. Νόμιζα θα ήταν πιο ειλικρινής στη διατύπωσή του. Είχαμε πει στο παρελθόν ότι υπήρχαν κάποιες επιφυλάξεις, όχι επιφυλάξεις, υπήρχαν αναστολές διορθώνων προγραμμάτων. Η χώρα η Γερμανία, λέτε ότι δεν έχει τέτοια προβλήματα, αλλά στην έκθεση αναφέρεται, λέτε 171 ε, χώρες, ότι είναι η Ιταλία, η Ισπανία κτλ. Στο 172 σημείο λέτε ότι χαίρεστε για τις αναστολές πληρωμών, αλλά δεν λέτε για ποιες χώρες. Σε ποιες χώρες είναι όλα αυτά. Εγώ πιστεύω ότι οι Ισπανοί πολίτες θα πρέπει να έχουν κάποια μεγαλύτερη διαφάνεια. Μας έχει, έχουμε βαρεθεί για τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά κύριε Πίπερ. Για τα θέματα των εσόδων, για το ΦΠΑ υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ Ισπανίας και Γερμανίας. Ε, 10 εκατομμύρια, 10 δισεκατομμύρια μάλλον, σε σχέση με την ίσπραξη ΦΠΑ σε βάρος της Γερμανίας. Εγώ τα κοίταξα όλα αυτά γιατί εσείς είπατε ότι έχει ληφθεί υπόψη αυτή η διαφορά για το ΦΠΑ, εγώ δεν το βλέπω πουθενά. Έχετε αυτό το κατάλογο που λέει Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Φιλανδία κτλ. Και οι επιφυλάξει είναι σαφεί, αλλά τα δύο μόνο προγράμματα τα οποία έχουν ανασταλεί στην ε, στην ε, περίοδο για την οποία είστε στις εισαγωγή περιλαμβάνουν και τη Γερμανία και εκεί δεν λέτε τίποτα. Οι πολίτε στην Ισπανία έχουν βαρεθεί λοιπόν να ακούνε τα ίδια και τα ίδια και δεν μπορώ να έχω ένα Γερμανό εισηγητή ο οποίο θέτει ένα αμφιβόλο την ε, εντιμότητα όλων εκτό από του Γερμανού. Δεν δέχομαι λοιπόν αυτά τα δύο μέτρα και δύο σταθμά τα οποία θέλετε εσείς να εφαρμοστεί. Και εσείς λέτε κύριε Σιωμέτα ότι θα είσαστε ο διαμεσολα διαμεσολαβητής, δεν είναι διαιτητής λέτε ότι είναι η Κομισιόν, αλλά πρέπει να παίξει το ρόλο του προπονητή. Όλοι αυτοί οι παίκτες θέλουν ένα καλό προπονητή που θα τους δείξει πώς θα κάνει καλά τη δουλειά του, γιατί δεν θέλουμε διαιτητές, θέλουμε κάποιον ο οποίος θα εκπαιδεύσει. Αυτό χρειάζεται όχι να λέτε ότι το πρόβλημα είναι στα κρατημέλη. Εσείς είστε υπεύθυνοι γιατί όλοι περιμένουμε από την Κομισιόν να φέρει σε πέρα στο καθήκον της που είναι η πρωτοβουλία και όχι να κακολογεί τους άλλους. Ευχαριστώ Η συνάδελφος Παναγιώτοβα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Θέλω καταρχήν να συγχαρώ τον εισηγητή για ό,τι έχει κάνει και για τις διαπιστώσεις του. Δυστυχώς, τρία συνεχή χρόνια η κοινή αγροτική πολιτική και η πολιτική συνοχής συνεχίζουν να σημειώνουν προβλήματα και λάθη ιδιαίτερα ως προς τις δημόσιες αγορές. Επομένως, συγχαίρω την Κομισιόν που προτείνει κυρώσεις και πρόστιμα πιο αυστηρά για χώρες που διαπράττουν αυτά τα λάθη. Ζητώ λοιπόν, ρωτώ λοιπόν τον Επίτροπο Σεμέτα, πιστεύετε ότι οι κανόνες, οι κυρώσεις, οι κανόνες εφαρμογής των κυρώσεων ή των προστήμων έχουν αποτέλεσμα, φέρνουν αποτέλεσμα Υπάρχει όντως πρόληψη, τα κράτη-μέλη είναι αυτή τη στιγμή, έχουν συνετιστεί, διορθώνονται όντως τα λάθη στη διαχείριση των ε, γνωσιακών ταμείων. Και τέλος, τι πιστεύετε, τι φρονείτε για την πρόταση του εισηγητή του κυρίου Πίπερ, δηλαδή τις δηλώσεις ή ειδικέ εκθέσεις αναφορές για τις χώρες που διαπράττουν τα περισσότερα λάθη. Έπειτα. μία παρατήρηση που αναφέρεται στην έκθεση, δηλαδή η παράγραφο 210, είναι μία απλή διόρθωση, δηλαδή 22 Ιανουαρίου πρέπει να λέει. Γιάν Μούλτερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρέπει να καθορίσουμε τη θέση μας, δεν το έχουμε ακόμη κάνει, μιλήσαμε πολύ, αλλά το βασικό πρόβλημα είναι ότι για 19 χρόνια δεν έχει ποτέ στηριχθεί η Κομισιόν από το Ελεκτικό Συνέδριο με εξαίρεση ένα έτος. Το Κοινοβούλιο πάντα χορηγούσε την απαλλαγή και δίναμε στην Κομισιόν, δείχναμε στην Κομισιόν την εμπιστοσύνη μας τουλάχιστον εν μέρη. Κάθε χρόνο δίνουμε την απαλλαγή, γίνονται πάντα υποσχέσεις και το αποτέλεσμα δεν υπάρχει. Υπάρχει λοιπόν εδώ ένα πρόβλημα. Όσο για τη σύγκριση της Κομισιόν με το διαιτητή ως προς την κίτρινη κάρτα, και ότι θα έπρεπε να την παίρνουν οι παίκτες. Ωραία σύγκριση, αλλά σύμφωνα με τις συνθήκες υπεύθυνοι είναι η Κομισιόν και εμείς δίνουμε απαλλαγή στην Κομισιόν και όχι στα κράτη-μέλη. Αν ήταν άλλες, άλλη η συνθήκη μπορεί να είχατε δίκιο, αλλά δεν είναι άλλη. Δέχομαι ότι το πρόβλημα έγκυται στα κράτη-μέλη και επομένω νομίζω ότι θα ήταν μια καλή ιδέα, ε, ότι είναι καλή ιδέα του εισηγητή με τις επιφυλάξεις. Έχω την εντύπωση όμως ότι η Κομισιόν αντιτίθεται στεναρά. 70% του προϋπολογισμού άρα δεν πρέπει να τύχει απαλλαγή. Καλό θα ήταν η Κομισιόν να μας πει γραπτός γιατί είναι κατά των επιφυλάξεων και ιδιαίτερα να μας εξηγήσει γιατί και η ίδια με τις δηλώσεις των γενικών διευθυντών έχει το δικαίωμα εκείνη να εκφράζει επιφυλάξεις. Ενώ εμείς λέει δεν έχουμε το δικαίωμα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αν μπορούσατε να μας στείλετε ένα σημείωμα γιατί είστε κατά των επιφυλάξεων και ταυτόχρονα γιατί εσείς μπορείτε να τις χρησιμοποιείτε και εμάς μας τις απαγορεύετε. Yeah, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ για τις παρεμβάσεις των συναδέλφων. Ευχαριστώ που τηρήσατε το χρόνο σας. Ο Επίτροπος να απαντήσει σύντομα. Το κύριο Σεμέτα. Για την τελευταία ερώτηση του Γιάν Μιούλντερ. Βεβαίως, βεβαίως. Θα σας στείλουμε γραπτό στα επιχειρήματά μας. Αναφέρθηκα στην επιστολή που θα στείλουμε στο Κοινοβούλιο και μπορούμε να αναφέρουμε γιατί θεωρούμε ότι οι πολιτικές επιφυλάξεις δεν είναι το σωστό μέσο. Οι επιφυλάξεις ή παρατηρήσεις που κάνουν οι Γενικές Διευθύνσεις είναι δυνατότητες διαχείρισης ε, που μεταφράζονται σε υποχρέωση ανάληψης πρωτοβουλειών για βελτίωση σε διαφόρους τομείς. Και ο ετήσιος χαρακτήρας των ελέγχων μας επιτρέπει να το κάνουμε αυτό. Συνολικά ωστόσο, σας καλώ να δείτε τα στοιχεία. Αν τα συγκρίνετε χρόνο το χρόνο, να δούμε το μέσο όρο της περίοδου 9-12, για παράδειγμα. Θα δείτε ότι το ποσοστό σφαλμάτων είναι 3,925. Ενώ ο μέσος όρος φέτος, τώρα που η Κομισιόν εισήγαγε ε, οικονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις ύψους 2% του προπολογισμού. Αυτό καταδεικνύει υψηλή απόδοση της Κομισιόν στην προστασία του ενωσιακού προϋπολογισμού. Παρακαλώ να το λάβετε υπόψη σας ε, όταν ε, αποτιμάτε την εργασία της Κομισιόν και πέρυσι. Πέρυσι το επίπεδο των ανακτήσεων και διορθώσεων αυξήθηκε ουσιοδός. Και τα επιχειρήματα ότι κάποιες από αυτές τις ε, διορθώσεις και τα λοιπά αφορούν την περίοδο 2000-2006 και δεν ανακλούν την ε, κατάσταση του 2012, δεν συμφωνώ με αυτό το επιχείρημα. Διότι αυτό αποδεικνύει, όπως είπε και η υφυπουργό ότι το πολιετές σύστημα ελέγχων μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Και αν ένα πρόβλημα αν ένα λάθος διαπραχθεί το 2012 θα διαπιστωθεί το 14 το λόγω των πολιετών ελέγχων. Έτσι λειτουργεί αυτό το σύστημα. Και κρίμα βέβαια που ανάλογα με τη συνθήκη το ελεκτικό συνέδριο κάνει τις εκθέσεις του ετησίως και δεν μπορεί έτσι να λάβει πλήρως υπόψη την ε, πολιτή φύση των ελέγχων και των διορθώσεων και ανακτήσεων του όλου συστήματος. Η κυρία Γιάννα Σέντερ είπε ότι πρέπει η Κομισιόν να είναι προπονητής. Ναι βεβαίως, προσπαθούμε να είμαστε καλοί προπονητές για τα κράτη-μέλη. Τους κάνουμε δηλαδή ασκήσεις δηλαδή τη δυνατότητα ανταλλαγής ε, βελτίστων πρακτικών. Το ανέφερε ο κ. Ρούμπικ για το προηγούμενο θέμα, ότι θα πρέπει η επιμόρφωση να βοηθήσει. Και πρέπει να πω ότι επενδύουμε πολλά στις δραστηριότητες επιμόρφωσης που αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη. Και αν θέλετε θα παρακαλέσω τις υπηρεσίες μου να σας δώσουν μια επισκόπηση των ε, πρωτοβουλειών κατάρτισης. Και τώρα με το νέο πολιτές πλαίσιο έχουμε τη δυνατότητα να επενδύσουμε παραπάνω για επιμόρφωση γιατί έχουν αλλάξει οι κανόνες και βεβαίως είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε Ούτως ώστε όσοι χειρίζονται αυτούς τους νέους κανόνες στα κράτη-μέλη να ξέρουν πώς πρέπει να τους χειριστούν. Τώρα, ο εισηγητής έδειξε συγκεκριμένα θέματα ότι πρέπει να γίνουν περισσότεροι έλεγχοι επί των δικαιούχων. Στα λεγόμενα πιο προβληματικά κράτη-μέλη. Η στρατηγική ελέγχων μας που εκπονείται αυτή τη στιγμή από τις υπηρεσίες μου θα βασίζεται στην αποτίμηση του κινδύνου. Δηλαδή, στα κράτη-μέλη όπου διαπιστώνουμε ε, την χείριστη απόδοση θα κάνουμε περισσότερους ελέγχους σε σχέση με τα κράτη-μέλη που τα πάνε καλύτερα. Και βεβαίως αυτό θα αφορά και τους ελέγχους των δικαιούχων. Ήδη συμβαίνει αυτό σε ορισμένους τομείς και πρόθεσή μας είναι να επεκταθεί. Η αντικατάσταση προγραμμάτων, αναφερθήκατε και σε αυτό. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο νέος κανονισμός δεν επιτρέπει αναδρομική αντικατάσταση. Αυτό είναι το θετικό από τον νέο κανονισμό. Αλλά είναι πολύ πρόσφατος αυτός ο κανονισμός. Αλλά ε, προβλέπει όμως παρόλα αυτά τη δυνατότητα λανθασμένα προγράμματα να αντικατασταθούν με καλύτερα προγράμματα εάν έχουν ε, διαπιστώσει τα ίδια τα κράτη-μέλη τα ασφάλματα και έχουν συμφωνήσει με τις δράσεις ελέγχου της Κομισιόν. Αυτό είναι ο κανόνας. Είσαστε μέλη, εσείς ευρωβουλευτές, στην Περιφερειακή Επιτροπή, στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Εσείς ψηφίσατε αυτά τα μέτρα, αυτές τις διατάξεις. Βδομάδες είναι, ή μάλλον μήνες, δύο μήνες που τα εγκρίνατε. Δεν καταλαβαίνω. Και το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε και για τις κυρώσει στη Γεωργία. Βεβαίως, να υπάρξουν καιρό στη Γεωργία. Αλλά συμφωνήσουμε επιτέλους. Εμείς και οι συνεισηγητές τι ακριβώς θέλουμε. Γιατί ξέρετε τους κανόνες που αποφασίζουμε μετά πρέπει να τους εφαρμόζουμε. Πλήρως. Και σε ορισμένα σημεία της έκθεσης αμφισβητείτε τις πολύ πρόσφατες ε, αποφάσεις σας επί νομοθετημάτων. Και εγώ δεν καταλαβαίνω μια τέτοια προσέγγιση. Όπως είπα και στην εισαγωγή μου, στα πλαίσια των κανόνων της νομοθεσίας, είτε είναι πρόσφατη είτε παλαιότερη. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά είμαστε απόλυτα δεδεθειμένοι να εφαρμόσουμε με μέγιστη αυστηρότητα τα μέτρα. Αλλά δεν μπορούμε ε, να κάνουμε περισσότερα από όσα προβλέπει η νομοθεσία. Να υπερβούμε την νομοθεσία. Αυτό σε μένα τουλάχιστον είναι σαφές. Τέλος. Όπως είπα και στην εισαγωγή μου, Είμαστε πλήρως ε, πρόθυμοι να συνεργαστούμε με την Επιτροπή σας για να συμβάλλουμε στη βελτίωση της διαχείρισης των ενωσιακών πόρων και σας καλώ την Επιτροπή σας και γενικότερα το Κοινοβούλιο να ξαναδούν αυτή την προσέγγιση πολιτικών επιφυλάξεων. Δεν νομίζουμε ότι είναι πιο κατάλληλη. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Δύο λεπτά ο Μάρκος Πίπερ για να τελειώσει η συζήτηση. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Σέντερ, θα ήθελα να σας πω. Υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να σας επιτρέψει να κοιτάξετε την ε, έκθεση. Αν το χρησιμοποιήσετε με προγράμματα αναζήτησης, ίσως δεν θα βρείτε αυτά τα οποία ε, θέλετε. Ε, οπότε διαβάστε ίσως πιο προσεκτικά την έκθεση. Λυπάμαι αν δεν λαμβάνετε υπόψη αρκετά το θέμα της Γερμανίας, αλλά δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό που είπατε για τη Γερμανία, ότι δεν εμφανίστε. Όλα τα κρατημέλη, σχεδόν όλα τα κρατημέλη αναφέρονται στην έκθεση. Αν κοιτάξετε λοιπόν την έκθεση, θα δείτε ότι υπάρχει και η Γερμανία. Δεν πρέπει λοιπόν να έχετε ανησυχίες ότι είναι κομματικού χαρακτήρα η έκθεση την οποία έχω υποβάλει για τα σχόλια των συναδέλφων. γιατί τους φιλελεύθερους και αυτά που είπανε ε, υπάρχει και σύμβη από τη δική μας πλευρά. Αν κατάλαβα καλά αυτά που είπε ο Ντέρεκ Βόμ για τις πολιτικές επιφυλάξεις και για τις ε, διεκδικήσεις που έχει διατυπώσει έχω τονίσει ότι εμείς είμαστε πάντα έτοιμοι να διευκρινίσουμε καλύτερα τι ακριβώς είναι αυτές οι πολιτικές προϋποθέσεις, πολιτικές επιφυλάξεις. Και κύριε Πίτροπε λοιπόν, ε, κατανοώ ότι θα μπορούσε κανείς να έχει παρανοήσεις, γιατί η πραγματικότητα, με διαβάσει κανεί την έκθεση προσεκτικά, είναι ότι εμεί υποστηρίζουμε πάντα το να έχει η Κομισιόν περισσότερε αρμοδιότητε εναντί των κρατών μελών και αυτό αναφέρεται κατ' επανάληψη. Λοιπόν, δεν θεωρούμε ότι εσεί είσαστε ο κακό σε αυτό το παιχνίδι. Δεν έχουμε τώρα πολύ χρόνο για να αντιμετωπίσουμε τι τροπολογίε. Θέλω να παροτρύνω τους ε, συναδέλφου τα μέλη τη Επιτροπή. να τις εξετάσουν για την Επιτροπή τώρα Περιφερειακών Θεμάτων. Εγώ έχω ψηφίσει πράγματι όπως ελέγχθη, αλλά επρόκειτο για ένα θέμα που είναι κάπως διαφορετικό. Εμείς βλέπουμε τα θέματα όχι από την ε, οπτική γωνία αυτών οι οποίοι είναι δικαιούχοι, αλλά με την οπτική γωνία αυτών που θέλουν να ελέγξουν την εφαρμογή αυτών των κονδυλίων και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον εισηγητή και όλους αυτούς οι οποίοι έλαβαν μέρος στη συζήτηση, λέει ο Πρόεδρος, και από τον κύριο Βέρχα από το Ελεκτικό Συνέδριο. Έχουμε κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν τώρα, για τα οποία θα πάρουμε ε, γραπτές απαντήσεις από τον κύριο Επίτροπο και μπορώ να κλείσω τη συνεδρία σήμερα και σας εύχομαι καλή επιστροφή.